Okay, colleagues, uh, could we start? We have a full uh, agenda. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλή δουλειά. Μεγάλη αίθουσα. Να κοιτάξουμε. Αν υπάρχουν ε, προσθήκες στην ημερήσια διάταξη, τα πρακτικά από την 29η Νοεμβρίου τα έχετε λάβει, υπάρχουν ε, προσθήκες. Να εγκρίνουμε λοιπόν τα πρακτικά και να κάνουμε τις ανακοινώσεις της Πρόεδρου στην ε, τελευταία συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρείου είχατε πει ότι στο Διευρυμένο Προεδρείο ΑΦΕΤ χρειάζεται να επιμείνουμε και να υπογραμμίσουμε ότι Ε, ότι θα αποφασίσουμε ορισμένα πράγματα μόνοι μας. Θέματα και ποιος θα αναλαμβάνει τις προσωρινές ε, εκθέσεις στην Επιτροπή των ε, Δικαιωμάτων και μετά η ΑΦΕΤ θα λαμβάνει τελική απόφαση σε κοινή συνεδρίαση με μένα βέβαια ο κύριος Μπροκ. Θα ορίζονται δε οι μελλοντικές πολιτικές. Η ατμόσφαιρα στο διευρυμένο Προεδρείο ΑΦΕΤ μου φάνηκε θετική. Πεστήριξαν όλες οι ομάδες ότι θα εργαστούμε περισσότερο, θα συνεργαστούμε και θα ενισχύσουμε και θα υποστηρίζουμε ο ένας τα προγράμματα, τις επιλογές του άλλου. Θα προσπαθήσουμε επίσης να αποφύγουμε επικάλυψη εργασιών κατά την επιλογή των διαφορών μελετών. Συνεδρίαση λοιπόν προβλέπεται στις δύο υποεπιτροπές ε, ε, κοινή στο Στρασβούργο. Με τις δύο υποεπιτροπές θα σας ενημερώσω. Επίσης είπαμε ότι θα επεξεργαστούμε ψήφισμα προς την ε, αποστολή αντιπροσωπείας για το Συμβούλιο των Δικαιωμάτων στη Γενέβη. Είχαμε μια επικοδομητική συνεδρίαση με κάποιους από τους συναδέλφους που θα πάνε εκεί, με τους αντιπροσώπους και έτσι την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε συνενετικό ψήφισμα με κάποιες τροπολογίες. Ψήφισμα το οποίο συνήθως είναι ταυτόσιμο από τη μια χρονιά στην άλλη, αλλά λόγω της ε, αραβικής Άνοιξη έχουμε προσθέσει μια-δύο παραγράφους για τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Επίσης ε, συνομίλησα με τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μάρτιν Σούλτσα. Θεώρησα ότι ήταν πολύ ε, ε, ευγενική χειρονομία του να δεχθεί να συναντήσει την πρόεδρο μιας υποεπιτροπής, έστω και με το θετικό πρόσημο δίπλα. Ε, Πάντω σκοπεύει να ανορθώσει από ό,τι φαίνεται το, την παρουσία του Κοινοβουλίου, να ενισχύσει το δημόσιο πρόσωπο του Κοινοβουλίου. Ε, πολλά ταξίδια δεν σκοπεύει να αναλάβει. Βέβαια θα πάει στην Κίνα και τη Ρωσία, αλλά δεδομένων και των οικονομικών περιορισμών μας βεβαίως ότι θα είναι περισσότερο ε, δραστήριος εδώ και όχι στο εξωτερικό. Ίσως λοιπόν το Σεπτέμβριο να έχουμε την ευκαιρία να τον συναντήσουμε να συναντήσουμε τον πρώην πρόεδρο για να μας πει και εκείνος τι έχει δει. Για το αντιπρόεδρος, ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ επανεξελέγει ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκτυο Ζαχάροφ. Έχει διεξαχθεί συνεδρία ομάδα εργασία για το χρηματοπιστωτικό μέσο, μέσο δημοκρατία και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ομάδα εργασίας της οποίας ηγείται η πρόεδρος της, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Δικαιωμάτων. Μέχρι στιγμή έχουμε σε τίσιο πρόγραμμα δράσης για το 2012 που έχει δηλαδή περισσότερο, μεγαλύτερο η χρηματοδότηση από ό,τι στο παρελθόν, αλλά όπως πάντα θα πρέπει να παρακολουθούμε ορισμένες εξελίξεις και η Άννα Γκόμες έχει ιδιαίτερα επιμείνει ως προς ορισμένες ε, εκλογικές αναμετρήσεις που θα πρέπει να σωματωθούν και στις σχετικές εκθέσεις. Επίσης, εχθές είχα μια συνάντηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα που μου έδωσε την ευκαιρία να συζητήσω για το πόσο δύσκολο είναι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε διάφορα κράτη ε, να εκφράσουν μέσα από την ιεραρχική τους δομή κάποιες επόψεις. Και πρέπει να πω ότι ήταν ε, μια εικόνα κάπως ε, ζωφερή. Ήταν όλο άντρες, ήταν όλα γκρίζα τα κουστούμια και γενικά ήταν μια πολύ ουδέτερη εικόνα αυτή που είχα μέχρι τώρα. Το, η, η καινούργια όμως εικόνα μου από τη χθεσινή επαφή με πολλές γυναίκες, πολλούς νέους, νέες γυναίκες, ε, χρώμα πολύ στη συνεδρίαση μου έδωσε άλλες ελπίδες. Φέρνουν λοιπόν την παρουσία μας. Και υπεγράψα και εγώ ότι είναι σημαντικό για μας να ε, παρακολουθούν τις συνεδριάσεις μας όταν είμαστε εδώ και όταν έρχεται να μας ομιλεί ο επικεφαλής αντιπροσωπείας. Επίσης εξελέγει νέος ύπατος εκπρόσωπος για ανθρώπινου ανθρώπινα ο κ. Μουτσνιέξη από τη Λετωνία πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Αδιαλαξίας από το Συμβουλίο της Ευρώπης και πιστεύω θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω σύντομα και να το προσκαλέσω στην προσοχή μου συνεδρί... στην προσοχή μας συνεδρίαση το... στο Στρασβούργο. Δεν θα συναντηθώ και με τον κύριο Χάμαρπερ και για να τον ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή μας. Ρωσία, Συρία. είχα δημοσιεύσει ε, ένα ανακοινωθέν ε, τύπου στις 4 Φεβρουαρίου όπου υπερθύμιζα στην ε, Ρωσία τις βασικές αρχές των ανθρωπινών δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης εν του ψηφίσματος για τη Συρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας που δεν ελευθεί υπόψη Πριν όμως το ανακοινωθέν τύπου είχα επίσης υπογραμμίσει ότι επικεντρωνόμαστε στην ε, ανάγκη οι ρωσικές αρχές να δηλώσουν ότι σέβονται τις ε, βασικές ελευθερίες και το δικαίωμα τους να έρχεσαν. Επίσης, σε μια συνάντηση με τον πρεσβευτή του Μαρόκου πριν από μερικές εβδομάδες, ε, έθιξα το ζήτημα της θανατικής ποινής που πικρεμόταν εις βάρος ενός πρώην πρωτοθλητού της πυγμαχίας υπεγράμμισε πόσο σημαντικό θα θεωρούνταν το να του χορηγηθεί χάρη από τον βασιλέα. Πράγμα το οποίο και συνέβη. Υπήρχαν και άλλε σχετικέ υποθέσει για τι οποίε όμω δεν έχω λάβει απάντηση. Επίση, έχω αποστείλει επιστολή σε αρχέ τη Ερυθρέα για την περίπτωση ενός ε, Σουηδού υπηκόου με το όνομα Νταβίτη Ισάκ που είναι ο πλέον ε, παλαιός κρατούμενος στις φυλακές εκεί και ζήτησα ο πρόεδρος Ασμάρα να ε, κοιτάξει την υπόθεσή του και να την παρακολουθήσει. σε αυτή η ήπια, η ήρεμη διπλωματία να βοηθήσει, πάντως πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Με τον Γκραφ Λάμστοφ πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας Ηνωμένων Εθνών, συμφωνήσαμε να ενημερώσουμε την ΑΦΕΤ για την επίσκεψή μας στη Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου. Πολλές φορές αλλάξαμε τις σημερομηνίες, αλλά δεν μπορέσαμε ακόμα να βρούμε κοινή συνεδρίαση. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι συμπροεδρεύσαμε τις αντιπροσωπείας η οποία είχε μέλη την κυρία Αντρικέινα και τον κύριο Σάλακ εκ μέρους της μαζί με μένα. Και συζητήσαμε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περισσότερες συζητήσεις μας, ιδιαίτερα την Μέση Ανατολή. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρεσβευτή του Ισραήλ και εκπρόσωπο των Παλαιστινίων. καθώς ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση είχε δοθεί στο πώς θα κρίνουν τα Ηνωμένα Έθνη η Γενική Συνέλευση το ε, αίτημα για αναγνώριση της κρατικής οντότητας της Παλαιστίνης. Ε, είχαμε επίσης ε, συναντήσεις με Λιβύα, Συρία, Αίγυπτο και με τον κύριο Κρίστοφερος για την ε, κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα που δεν ε, μπορώ να σας εκθέσω σε κάθε λεπτομέρεια αλλά πάντως θεωρεί εκείνος ότι η Αραβική Άνοιξη δεν προσέφερε πολλά πράγματα στην ε, αναζήτηση πολιτικής λύσης αλλά ούτε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Την Δυτική Σαχάρα την έχουμε βάλει στο πρόγραμμα μας για το πρώτο ήμιση του έτους και θα κοιτάξω αν μαζί με την ΑΦΕΤ και τον κύριο Μπρότ μπορούσαμε να οργανώσουμε μια κοινή συνεδρίαση και όπως είπε ο Κρίστοφερ Ρος είναι διατεθειμένος να έρθει αλλά καθώς δεν είχε δεχθεί πέρσι την πρόσκληση της ΑΦΕΤ θα πρέπει να δείξουμε μια ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επίσκεψή του εδώ. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα μάθαμε από τον επικεφαλής της ε, Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας εκεί ότι επηρεάζει η Αραβική Άνοιξη της, ε, το πνεύμα της συνεδριάσης και τις ψηφοφορίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αλλάζουν ε, τρόπο τοποθέτηση κατά τι ψηφοφορίε σε ορισμένε αραβικέ χώρε. Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, γίνεται μια καλύτερη προσπάθεια για ενσωμάτωση στο πλαίσιο των Εθνών του ζητήματο προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ταυτόχρονα λοιπόν, Νοέμβριο πάντα, διαπιστώσαμε ω ε, θετικό το γεγονό ότι ετοιμαζόταν ψήφισμα για τη Συρία, έστω κάπως απαιτητικό, που επεδίωκαν να περάσει. Και, εν πάση περιπτώσει, έμεινε μέχρι εκεί όμως η υπόθεση του ψηφίσματος, δεν έφτασε μέχρι το Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί βέβαια ταυτόχρονα υπήρχε και το αίτημα της ε, καταγγελίας ε, των σοβαρών ε, εγκλημάτων πολέμου που έκρινε το ψήφισμα αυτό και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Πολέμου, πράγμα το οποίο βεβαίως δεν αποφασίστηκε. Εν τέλει δεν ενεκρίθη. Επίσης είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ειδικό συζητητής, ειδικό ε, μηχανισμός για το Ιράν, πράγμα το οποίο μάλλον δεν θα επιτευχθεί. Και επίσης ε, για την ε, οικουμενική περιοδική έκθεση μας είπαν ότι οι κυβερνήσει δέχονται περισσότερες επικρίσεις και δέχονται επίσης να εκτίθενται στην κριτική από άλλες χώρε και γενικώ κρίνουν θετική την θετικές τις επιδόσεις αυτού του γύρου οικουμενικής αξιολόγησης. Τώρα στο δεύτερο γύρο που βρισκόμαστε θα πρέπει να δούμε αν όντω υλοποιούνται τα υπεσχημένα εκ μέρους των κρατών για να έχουμε μια πιο επακριβή κρίση, αν δηλαδή αυτή η οικουμενική κρίση μπορεί να φέρει κάποιες ουσιαστικές αλλαγές. Εν γέννη, κρίνω καλό το ότι έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΑΦΕΤ και της, ε, και της Αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Εθνών και της Επιτροπής για τα, πολιτικά, για, τις, για τα Δικαιώματα. Ε, ο κύριος Γκραφ ε, Τσουλάνσδορφ ήταν πολύ συνεργάσιμος, μπόρεσα και εγώ να συζητήσω μαζί του διάφορα θέματα. Οπότε φαίνεται ο Γκραφ Λάνστορφ θα ε, αναφερθεί στη ε, ΑΦΕΤ στις 29 Φεβρουαρίου όπου εγώ θα είμαι επικεφαλής αντιπροσωπείας θα βρίσκομαι στη Βιρμανία και άρα θα παρακαλέσω την κυρία Αντρικέινε να είναι παρούσα στην ε, συνεδρίαση Γκραφ Λάντστορφ και ΑΦΕΤ για να μας ενημερώσει μετά. Αυτά ως προς ανακοινώσεις της Προέδρου. Περνάμε τώρα στο πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης. ενημέρωση και συζήτηση από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την κοινή ανακοίνωση ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Οπότε Παρακολουθούμε όλοι αυτή την έκθεση. Θα συζητήσουμε την ανακοίνωση της κυρίας Άστον, ε, ανακοίνωση του Δεκεμβρίου, η οποία αποτελεί τη βάση για τη συζήτησή μας πριν ε, βεβαίως δημοσιευτεί η έκθεση αυτή ανησυχούσαμε για την διαδικασία γιατί εάν ήταν αυτή η τελευταία λέξη στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα μας ικανοποιούσε το ότι εμείς δεν είχαμε χρόνο λεπτομερός να συνεισφέρουμε στη συζήτηση κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Αποστήλαμε λοιπόν κάποια συνεισφορά ως διευρυμένο Προεδρείο και τέλη Νοεμβρίου νομίζω πως αυτό το βλέπουμε ως μια αφετηρία κατά το οποίο καλωσορίζουμε Ανέφερα κάποια πράγματα λοιπόν, το ότι είναι σημαντικό για εμάς και τώρα καλωσορίζουμε το ότι έχουμε περισσότερο χρόνο και το ότι και τα κράτη-μέλη ξεκινούν να συζητάνε πιο δυναμικά από την πριν επί της ουσίας και το ότι τώρα από ό,τι καταλαβαίνω θέλουν μια συνολική προσέγγιση και ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα βοηθήσει και να επιτηρήσουμε την κατάσταση. Αυτά μέχρι στιγμή και έχουμε και το προηγούμενο βεβαίω σημείο στην διάταξη όταν ε, είχαμε συζητήσει την ετήσια έκθεση του 2010 είχαμε αποφασίσει πως η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιέχει και κάποια πράγματα για την έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε θα το δούμε από διάφορες πτυχές. Σήμερα δε το πρωί μόλις αποφασίσαμε πως η έκθεση του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πάει στους πράσινους, στον κύριο Ταβάρες και νομίζω πως τώρα τίποτα δεν μας εμποδίζει να μπούμε στις λεπτομέρειες και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Ποπόφσκι που ασχολείται από πλευράς υπηρεσίας εξωτερικής δράσης με το θέμα και το προωθεί και θα ξεκινήσει παρουσιάζοντάς μας το πόσο έχουν προχωρήσει τα πράγματα και η συζήτηση για την ε, εξέταση των Να σας πενθυμίσω επίσης πως κάναμε την πρόταση στο τέλος αυτής της διαδικασίας αναθεώρησης όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία είτε είναι δήλωση ή κάτι ανάλογο να τονίσουν το πόσο σημαντικά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα δούμε τι θα γίνει ως προς αυτό. Είναι θετικά αυτά τα πράγματα. Το έθεσα και στη συζήτηση με την Υπουργό Εξωτερικών της Δανίας. Δεν είναι εναντίον, αλλά οπωσδήποτε κάποια κράτη-μέλη δεν είναι κατά, η ΜΚΟ δεν είναι κατά γιατί θα ενισχυθούν, αλλά το σημαντικό είναι τώρα να δούμε πώς θα το επιτύχουμε. Και οπωσδήποτε να αποκτήσει μια ουσία η υπόθεση και να υπογραμμίσουμε την δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το είπαμε και στον πρόεδρο Σούλτς πως καλό θα ήταν και έχουμε δυόμιση χρόνια ακόμα στην θητεία βεβαίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ θα ήθελα να γίνει αυτό εντός της Προεδρίας της Δανίας. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Ποπόφσκι και να μας ενημερώσει για το που έχει φτάσει στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα. Με συγχωρείτε που είμαι άντρας και γκρίζος αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είπατε πράγματι πως είναι η αρχή μιας διαδικασίας αλλά ξέρετε πως υπάρχει ένα ιστορικό στη διαδικασία και δίκαιο. Νομίζω μπορούμε να πούμε πως δεν ήταν ε, εύκολα τα πράγματα όσον αφορά την πρώτη αυτή αναθεώρηση της πολιτικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θεωρήσαμε πως καλό ήταν να έχουμε γερά θεμέλια πριν αρχίσουμε να χτίζουμε και Οπωσδήποτε ο χρόνος που αφιερώσαμε στις απόψεις των ενδιαφερομένων δεν σπαταλήθηκε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εμπλακεί από νωρίς ε, στην διαδικασία αυτή. Ε, ο πρόεδρος του ή άλλως τον Ιούλιο του 2010 ήταν και στο 12ο φόρουμ με τις ΜΚΟ και στην Υποεπιτροπή και με μονομένους βουλευτές βεβαίως μετά είχαμε διάφορες συναντήσεις πέρα βεβαίως από τις τακτικές εμφανίσεις της ΙΠΑ της εκπροσώπου ε, που τελευταία φορά ήρθε τον Δεκέμβριο. Είμαι σίγουρος πως ε, θα γνωρίζετε βεβαίως το περιεχόμενο της κοινή ανακοίνωσης να υπενθυμίσω τα βασικά σημεία αφού έγινε ένας απολογισμός λοιπόν του πλαισίου της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποφασίστηκε μια αντίδραση σε τέσσερα μέρη. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής, δηλαδή μια συγκεκριμένη προσέγγιση που θα σχετίζεται με κάποιες εκστρατείες, με βάση κάποια θέματα που έθεσε η κάθε άστον ε, μεταρρύθμιση δικαιοσύνης, δικαιώματα των γυναικών και δικαιώματα των ε, παιδιών για να έχουμε μια νέα προσέγγιση στην πολιτική γειτονία και παραπέρα και βεβαίως εμπλοκή με την κοινωνία των πολιτών δεύτερων. Στοχεύουμε να έχουμε μια συνολική συνοχή στην πολιτική μας για να έχουμε μια συνοχή σε διάφορους τομείς της πολιτικής που συνήθως βλέπουμε απομονωμένους. Εμπόριο, αντιμετώπιση των κρίσεων, ελευθερία, δικαιοσύνη, αντιτρομοκρατία. Δανειστήκαμε λοιπόν κάποια πράγματα από την έκθεση του Κόφι Ανάν λέγοντας πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια και δεν θα υπάρξει τίποτα από τα δύο χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν λοιπόν τα μέσα τα οποία είναι ε, οι ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες συμφωνίες. Κατόπιν βεβαίως υπάρχουν οι ισχυρές εταιρικές σχέσεις διμερείς ή πολυμερείς ε, όσον αφορά τους όρους ε, των διεθνών αυτών σχέσεων και τέλος δίνουμε μεγάλο βάρος στο να φροντίσουμε όλες μας οι προσπάθειες σε όλο το φάσμα της πολιτικής να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι με το να πάμε σε μια ομάδα εργασίας που θα βασίζεται στις Βρυξέλλες που σιγά σιγά υλοποιείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της επικοινωνίας των ζητημάτων αυτών. Δεν θα αλλάξει τίποτα βεβαίως εάν δεν βρούμε ένα τρόπο να εφαρμοστούν αυτές οι ιδέες. Όπως λέει η ανακοίνωση, αυτό σκοπεύει να αποτελέσει συνεισφορά στην συζήτηση που υπάρχει και αναζητά απόψεις για πιθανές δράσεις και επιλογές και επόμενο βήμα θα είναι μέσω των διοργανικών συζητήσεων να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και είναι σαφές πως ε, το Κοινοβούλιο έχει ήδη σημαδέψει την διαδικασία. Όπως ακούσατε η κάθε άστον όρισε έναν ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να αυξηθεί και το προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ήδη έχουμε τις πρώτες κινήσεις. Την τρίτη αυτής της εβδομάδας έλαβε χώρα μια πρώτη συζήτηση στο Συμβούλιο στην Επιτροπή, ε, στην Πολιτική Επιτροπή Ασφαλείας. Εκφράστηκαν λοιπόν διάφορες ε, ιδέες για το τι καθήκοντα θα μπορούσε να έχει ο ειδικό αυτός απεσταλμένος και έχουμε άρα μια εντολή η οποία κατά βάση θα αφορά τον έξω κόσμο να αυξήσει δηλαδή την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει πρόσβαση υψηλού επίπεδου σε ξένες κυβερνήσεις και στο διεθνές πλαίσιο. Εξυπακούεται πως ε, ο αυτός ο απεσταλμένος βεβαίω θα πρέπει να μπορεί να εντάσσεται στις υφιστάμενες δομές της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και να μην κάνουμε δύο φορές την ίδια δουλειά. και βεβαίως έχει ζωτικής, ε, ζωτική σημασία το έργο αυτό και θα πρέπει βεβαίω να δούμε και την νομική πτυχή της εντολής ε, που πιθανώς θα έχει καθώς για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ορίσει ε, ειδικό πρόσωπο για ένα ζήτημα θεματικό συγκεκριμένο γιατί πάντα επικεντρωνόμαστε με γεωγραφικό τρόπο και όχι με τρόπο θεματικό Υπήρχε βεβαίως, υπήρχαν ειδικοί εκπρόσωποι του τότε, είπα του εκπροσώπου του Χαβιέ Σολάνα, η κυρία που κάθεται στα αριστερά μου. Οπότε ε, πρέπει να δούμε τι γράφει η συνθήκη, πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά και από νομική σκοπιά πρέπει να συνεργαστούμε με την Κομισιόν για να φροντίσουμε πως η εντολή θα ε, στέκει νομικά καθώς τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ξεφεύγουν από το πεδίο της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Επίσης, η Πολιτική Επιτροπή συζήτησε τη δυνατότητα ενός μελλοντικού σχεδίου δράσης στη φάση εφαρμογής της ε, εξέτασης αυτής των πραγμάτων. Νομίζω πως υπήρχε μια θετική ε, αντιμετώπιση, όχι ομοφωνία, είναι νωρίς ακόμα, αλλά αρκετά θετική αντιμετώπιση, οπότε η υπηρεσία μας άρχισε να σκέφτεται τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει το σχέδιο δράσης ε, και θα υποβάλουμε προτάσεις τις ερχόμενες ε, εβδομάδες. Κάποια από τα κράτη-μέλη επίσης ζήτησαν ε, ένα πολιτικό έγγραφο τώρα το εάν θα είναι δήλωση συμπεράσματα συμβουλίου θα το δούμε Πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή πριν το επόμενο βήμα μας για το πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μην επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα σε πολλά έγγραφα, γιατί βεβαίως θέμα να προσανατολιστούμε στη δράση. Βεβαίω ακούμε όλε αυτέ τι ιδέε και σημείωσα αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπίλερ για το Κοινοβούλιο. Και πράγματι θέλουμε η δουλειά του Κοινοβουλίου, η δική σας η δουλειά για την έκθεση αυτή να συνεισφέρει σε αυτό το οποίο γίνεται στο Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε μια κοινή πλατφόρμα όλων των θεσμικών οργάνων. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας και πολλά κρατημέλη ε, επίσης το ίδιο σκέφτονται. Υπάρχει λοιπόν μια καλή αφετηρία. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα μας ενθάρρυναν τα κράτη-μέλη και είναι και η δική μας η φιλοδοξία να οριστικοποιήσουμε την συνέχεια που θα δοθεί και βεβαίως για το σχέδιο δράση και για την εντολή του ειδικού απεσταλμένου. Όσον αφορά την διαδικασία, βεβαίως ε, θα υπάρξει μία συζήτηση των Υπουργών στην Κοπενχάγη νομίζω αρχές ε, Μαρτίου 8 και 9 Μαρτίου όπου η καθιάστον ε, πρότεινε μία συζήτηση σε επίπεδο Υπουργών Βεβαίω μια γενική συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα επί τη ευκαιρία και νομίζω πως ε, το δέχτηκαν πάρα πολύ θετικά οι Υπουργοί. Όσον αφορά βέβαια και την επιστολή που παραδοσιακά αποστέλει κάθε άστον πριν από τα άτυπα συμβούλια. Και βεβαίω τώρα θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για το πώς βλέπετε τα επόμενα βήματα για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το έργο της υπηρεσίας μας για το ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί στην ανακοίνωση και να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα στην αρχή πως η ανακοίνωση ήταν ένα πρώτο βήμα ήταν η ευκαιρία για τον ύπατο εκπρόσωπο την ύπατη εκπρόσωπο βεβαίως να παρουσιάσει τις απόψεις της για να συνεισφέρει στην αναθεώρηση αυτή του στήματος θα είναι μια κοινή προσπάθεια όλων των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστούμε κύριε Ποπόφσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Πριν δώσω το λόγο στον David Nichols από την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Είπατε κύριε Ποπόφσκι ότι το χρονοδιάγραμμά μας είναι μέχρι τον Ιούνιο. Ε, αποφασίσαμε με την γραμματεία για τον ορισμό ενός εισηγητή και ίσως εγκρίνουμε την έκθεση αυτή αναθεώρηση στην ενδιάμεση έκθεση μέχρι τον Ιούνιο. Γι' αυτό θα, έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ο Ντέιβιτ Νίκολς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να ε, αποτανθώ στην Επιτροπή σας μετά από την επανεκλογή σας και ε, προσδοκώ με μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ως προς την ανακοίνωση λοιπόν, πολύ εργαστήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και συμφωνούμε με αυτά που προείπε ο κύριος Ποπόφσκι ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η διαδικασία κατά την τελευταία διετία και ήταν άκρος απογοητευτική σε πολλά σημεία. Γι' αυτό είναι και ενθαρρυντικό αλλά και ανησυχητικό το ότι έχουμε ένα έγγραφο επιτάπητο στην αρχή μιας νέας διαδικασίας γιατί δεν έχουμε ολοκληρωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα. Πρόκειται για ένα έγγραφο, το οποίο θίγει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντά υπό την παρούσα του μορφή. Γι' αυτό ελπίζω ότι κατά τους επόμενους έξι μήνες θα συζητήσουμε τις απαντήσεις με όλα τα θεσμικά όργανα, με το Κοινοβούλιο και με την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει όμως ε, με σπουδή να δοθούν απαντήσεις γιατί ενώ συζητάμε για την αναθεώρηση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα τελευταία δυόμιση χρόνια, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει ήδη εφαρμοστεί αυτή η πολιτική. Και αυτό αφορά και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να έχουμε μια πολιτική η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί στο τέλος της ε, Προεδρίας της Δανίας. Η ανακοίνωση που έχουμε λοιπόν φύγει πολλά περισσότερα ερωτήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ στο έγγραφό μας πέρσι τον Οκτώβριο που ενήχε οκτώ σημεία έτσι ώστε να έχουμε μια σωστή πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θεωρούμε ότι η διαδικασία αναθεώρησης θα πρέπει να είναι ε, ολοκληρωμένη. Αν δούμε αυτά τα οκτώ σημεία, βλέπουμε ότι έγινε κάποια πρόοδος, αλλά θα ήθελα να δούμε ορισμένα από αυτά τα σημεία. Μιλήσαμε για την στρατηγική αυτή ως προς τις ανθρώπινες αξίες και δικαιώματα με βάση διεθνή πρότυπα. Τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε μία επιδείνωση ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα θεσμικά όργανα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή βρισκόμαστε μακριά από καθολικές αξίες και μιλάμε για ευρωπαϊκές καθαρά σε αυτή την ανακοίνωση καθίσταται σαφές ότι μιλάμε για, το αδιέρετο, για τον αδιέρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τον αναφέρετο χαρακτήρα τους. Επίσης, ασχοληθήκαμε με θέματα εσωτερικής-εξωτερικής συνοχής. Αυτό που είδαμε την ανακοίνωση αφορά μία αλλαγή 360 μοιρών. Όπως και η διεθνής αμνηστία είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει συνοχή ως προς την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Η ανακοίνωση αυτή για πρώτη φορά ασχολείται σοβαρά με αυτό το ζήτημα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Κατά τη Βελγική Προεδρία αναλήφθησαν πολλές πρωτοβουλίες και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο λαμβάνεται υπόψη σοβαρά. Οι ερωτήσεις, τα ερωτήματα ενυπάρχουν στην ανακοίνωση, αλλά όχι οι απαντήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τους επόμενους μήνες πώς μπορούμε να βρούμε ένα μηχανισμό που να ασχολείται ουσιαστικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιμετώπιση τους. Ένα άλλο θέμα που θίγουμε στο έγγραφό μας μιλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο όλων των μελημάτων μας. Αυτό αναφέρεται και στην ανακοίνωση, αλλά δεν ξέρουμε έμπρακτα πώς θα εφαρμοστεί. Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν στην ανακοίνωση είναι αυτή η σύγχυση ως προς τον επιμερισμό καθηκόντων. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για άτομα για πρόσωπα τα οποία δεν εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα θίγεται στην ανακοίνωση, αλλά δεν υπάρχουν απαντήσεις ακόμα. Δεν ξέρουμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε άλλους τομείς. Μιλάμε λοιπόν για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής και βλέπουμε ότι ως προς την εφαρμογή του πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, υπολοιπόμαστε κατά πολύ. Ελπίζουμε ότι αυτό το θέμα θα το αντιμετωπίσει το Συμβούλιο εφεξής στην απάντησή του ως προς την ανακοίνωση, μίλησε για το ρόλο των κρατών μελών και πιστεύω ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε και να δοθεί μια απάντηση κατά το επόμενο εξάμεινο. Το πέμπτο θέμα που θίξαμε αφορά την κατάρτιση για το προσωπικό καθώς και την αποτελεσματικότητα και απόδοσή μας και του διπλωματικού προσωπικού της ΕΙΕΔ. Η εκπαίδευση αναφέρεται στην ανακοίνωση, αλλά δεν μιλάμε για τον υποχρεωτικό της χαρακτήρα για την ΕΙΕΔ, καθώς και για τους επικεφαλείς ε, αντιπροσωπιών. Άρα δεν μιλάμε για μία συνεχή αξιολόγηση σε προσωπική βάση. Το έκτο σημείο που θίξαμε αφορά την διαφάνεια και τη ε, λογοδοσία, ιδιαίτερα ως προς την εταιρική μας σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει καλή επικοινωνία και ξανασκεφτήκαμε πολλά ζητήματα. Μετά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική πέρσι ως προς το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών Πρόκειται για έναν ισότιμο εταίρο. Υπάρχουν δυνατότητες διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, αλλά δεν αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της λήψης αποφάσεων. Συντάξαμε ένα έγγραφο λοιπόν για τις ε, διαβουλεύσεις. Το στείλαμε στη Βαρόνη Άστον στα τέλη κατά τα τέλη του 2010 για να δούμε πώς θα οριστικοποιηθεί αυτή η αναθεώρηση. Το έβδομο σημείο αφορά την ύπατη εκπρόσωπο και το διορισμό ενός ειδικού ε, εκπροσώπου μέχρι το τέλος της ε, Δανικής Προεδρίας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να προωθηθεί. Επίσης αποστήλαμε μία επιστολή για τον ιδεατό χαρακτήρα αυτής της εντολής και για το ρόλο μας ενδοκινοτικά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 8ο σημείο αφορά την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου ως προς τις υποδομές ε, που δημιουργούνται. Αυτό δεν ε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Περιμένουμε ε, μία απόκριση από το Συμβούλιο. Ήδη κατά την Αυστριακή Προεδρία είχε πρωτοθυγεί το θέμα και μας ενδιαφέρει να δούμε το θέμα αυτού του χειρισμού περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το έγγραφο δεν ετέθησε εφαρμογή και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει θέση. Το τελευταίο θέμα αφορά την συλλογική συμμετοχή των θεσμικών οργάνων. Δεν μιλάμε μόνο για την ΕΙΕΒ ή για ένα έγγραφο, αλλά μια συνολική προσέγγιση. Προσπαθούμε να εξεύουμε τρόπους έτσι ώστε να ε, υποβληθεί ένα κοινό έγγραφο μέχρι το τέλος της Προεδρίας, της τρέχουσας ε, Προεδρίας, σε επίπεδο ΕΙΕΔ, Επιτροπής και Συμβουλίου. Έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε μία πραγματική πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κύριε Νίκολς και ευχαριστούμε και ολόκληρο το δίκτυο διότι παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς αυτή τη διαδικασία διότι οι διάφορες ΜΚΟ ε, μέσα σε αυτή την περίοδο έχουν ωφεληθεί από τις συστάσεις σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ταβάρη, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον κύριο Ποπόφ, ευχαριστώ τους κυρίους Παπάς και Νίκολς. Προσδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτό το έγγραφο και θεωρούμε ότι ε, εμπεριέχει ενδιαφέρουσες ιδέες που θα θέλαμε να αναπτυχθούν ε, περαιτέρω από εμάς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ε, ευρύτερη συζήτηση για το ποια θα είναι η μεθοδολογία μας και η εφαρμογή των πολιτικών μας επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ ομιλώ ως ε, εισηγητής από πλευράς των Πρασίνων και θα ήθελα να πω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες προσδίδουν μεγάλη σημασία στην έκθεση αυτή. Ήδη το Κοινοβούλιο ασχολείται με τις στρατηγικές ε, επιπτώσεις αυτού του εγγράφου θα το δούμε και με τον κύριο Χάουιτ. Όπως ξέρετε έχουμε μία ε, μακροχρόνια παράδοση ως κοινοβούλιο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω δεν υπερβάλλω αν πω ότι το κοινοβούλιο μας διαδραμάτισε μοναδικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήμασταν ιδιαίτερα ε, δημιουργικοί σε αυτόν τον τομέα και νομίζω ότι αυτό αφορά όλες τις ε, πολιτικές ομάδες και την απάντηση στην ανακοίνωση με μια έκθεση του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να πω τα εξή. Όπως είπε και η Πρόεδρος, αυτό είναι σημείο εκκίνησης. Και εδώ ανακύπτουν τα πραγματικά ζητήματα, θέματα μεθοδολογίας, ε, θέματα ως προς το πρόγραμμα δράσης. Ο, ο κύριοι Ποπόφσκι και Νίκολς θίξαν ορισμένα επιμέρους ζητήματα και αυτό που έχει σημασία είναι πώς ε, μπορούμε να προωθήσουμε διαπραγματεύσεις και να δούμε πώς θα διαρθρώσουμε αυτές τις διαβουλεύσεις έτσι ώστε να έχουμε ε, μία αντικειμενική πληροφόρηση. Εμείς ε, είμαστε ένα πολιτικό σώμα, όχι διπλωματικό. και οι αντιλήψεις μας θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες πληροφορίες και σε μια πολύ καλή συνεργασία με την ΕΙΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν πρόσφατα θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία που θεωρώ ότι έχουν σημασία και θα πρέπει να μας απασχολήσουν ακόμα και αν επέλθουν αλλαγές, όπως είδαμε ε, ότι συνέβη με την Αραβική Άνοιξη, αλλά πολλά άλλαξαν και εντός Ευρώπης. Είχαμε θεσμικές αλλαγές με τη συνθήκη της Λισαβόνας, και ως απότοκο της ε, κρίσης ως προς τα μέτρα που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Ίσως αυτό να μην σχετίζεται άμεσα με την πολιτική περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, διότι ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανά τον κόσμο πολύ εξαρτώνται από τις θέσεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδαμε σε ορισμένα κράτη-μέλη ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση από αυτή την κρίση ως προς την οικονομική υποστήριξη, πολιτικό συντονισμό και διάλογο με τρίτες χώρες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή πώς να είναι ευέλικτη, πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική εν καιρό κρίσης και πώς ε, να ενισχύσουμε τους εταίρους μας ανά τον κόσμο, οι οποίοι είναι ενισχυμένοι αλλά δεν έχουν προωθήσει τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε σε θέση να το πούμε αυτό, γιατί η Ευρώπη θα είναι πιο αξιόπιστη αν αρχίσουμε από τα του οίκου μας, δηλαδή να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη-μέλη μας, κάτι το οποίο γίνεται και αν αρχίσουμε εκ των έσω βλέπουμε πώς βρούν, ας πούμε και οι επιχειρήσεις μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να δούμε θέματα εταιρικής ευθύνης που πολλές φορές ε, υποσκάπτει τη, τη δράση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τις συζητήσεις αυτού του εγγράφου τα θεσμικά όργανα κινούνται προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής ε, δήλωσης που έχει μεγάλη σημασία για όλα αυτά τα ζητήματα και για το πολιτικό μας σκέπτεσθε έτσι ώστε να εγκρίνουμε ένα έγγραφο το οποίο να έχει ιδιαίτερα ισχυρό περιεχόμενο από πολιτικής πλευράς και να είμαστε και επικοδομητικοί και παραγωγικοί ως προς το περιεχόμενο. Δεν πρόκειται για πολιτική δήλωση απλώς, αλλά για ένα έγγραφο με σαφές περιεχόμενο. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, να εργαστούμε υπό αυτούς τους όρους και είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε ιδιαίτερα παραγωγική από όλες τις ε, πλευρές του πολιτικού φάσματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Χάουιτ. Ευχαριστώ πολύ. Και καλώς ήρθατε για δεύτερη φορά στην Επιτροπή μας να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Με μεγάλη χαρά συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια. Έχουμε βέβαια επικρίνει πολλέ φορέ στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα ήθελα ωστόσο να σα ε, καθησυχάσω και να πω ότι και η κυρία και εγώ και άλλοι συνάδελφοι όπως ε, και οι εκθέσεις μας όπως η έκθεση για τα ε, για το Συμβούλιο Εθνικών Δικαιωμάτων που θα, περάσουν από, θα περάσει από την άλλη μέρα την επόμενη εβδομάδα, παρακολουθούν πάντα, παρακολουθούμε πάντοτε την ίδια γραμμή και έχουμε μια σταθερά, ε, σταθερή συμπεριφορά αντί τη Επιτροπή των Εξωτερικών Σχέσεων ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σα διαβεβαιώσω ότι είναι σαφέ το μήνυμα που θα πρέπει να αποστείλετε προ το Κοινοβούλιο ολόκληρο. Καλώς ήρθατε όσο ακούστηκαν από τον κύριο Παπόφσκι σήμερα ως προς τις αξίες και αρχές όντως είναι πολύ σαφές και καλό το κείμενο της Βαρόνης Άστον. Όταν μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ομολογήσουμε πως δεν είμαστε πάντοτε προσεκτικοί όσο θα έπρεπε στην προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων και το ανθρωπιστικό, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. αυτό λοιπόν έχει ε, αυτό έχει καταγραφεί στο κείμενο και πρέπει να πω ότι οι προθέσεις της υπάτης ε, εκπροσώπου της κυρίας Άστον ε, για μια πιο ουσιαστική διεθνή παρουσία και πολιτική με βρίσκουν σύμφωνο. Ξέρω ότι αυτή είναι η δική της πρόθεση, να μην περιοριστεί μόνο σε δηλώσεις, αλλά να προχωρήσει περισσότερο στην πράξη. Και πολύ καλά πράττει. Θα ήθελα επίσης να στηρίξω ρητά τα όσα είπε η κυρία Άστον στην Ολομέλεια. Το Δεκέμβριο. Ότι έχει με πολύ μεγάλη προσοχή παρακολουθήσει και αναλογιστεί τα όσα έχουν υποθεί και σχεδιαστεί ως προς την εντολή της ύπατης εκπροσώπου. Πρέπει λοιπόν ο έπατος εκπρόσωπος να είναι και ειδικό ε, βεβαίως ε, στην ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα και εκείνο που θα κληθεί να εκπροσωπήσει την υπατή εκπρόσωπο επίσης πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη στον τομέα των ανθρωπινών δικαιωμάτων και να μπορεί να διαπραγματεύεται για τα θέματα αυτά. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία έχουμε επισημάνει και στο Κοινοβούλιο και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για χρόνια και είναι όντως πολύ θετικό για μας το ότι έχουν επιτέλους ε, υιοθετηθεί αυτά που ζητούσαμε τόσα χρόνια. Βέβαια, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν είναι τόσο ενθουσιώδεις γιατί έχουν ε, διαπιστώσει ότι κάποια, από τη, κάποια κομμάτια της θεματολογίας που θέλουν να προβάλλουν δεν έχουν συμπεριληφθεί στην εντολή. Αλλά το βασικό είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα στον κόσμο, θέλουμε να φέρουμε ουσιαστικέ αλλαγέ. Και ίσως θα μπορούσαμε αυτό να το καταφέρουμε ε, με μία ε, μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων και εναλλαγή στα θέματα, όπως πράττουν άλλες χώρες, όπως η Ρώσοι, και θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς. Κάποιες από τις ε, ιδέες στην υλοποίηση των προτάσεων νομίζω θα πρέπει να ε, τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Γιατί εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν και πρέπει να γίνει μια συζήτηση πιο ουσιαστική. όπως άλλωστε εκφράζεται και η επιθυμία από διάφορες πλευρές. Στην Ολομέλη επίσης έχουμε μιλήσει για τους διαλόγους των ανθρωπινών δικαιωμάτων που είχα αποκαλέσει αποτυχημένους μηχανισμούς. Αυτό σε μια προσπάθεια να τραβήξω την προσοχή σας ε, στο γεγονός ότι λειτουργούν χειρότερα αυτοί οι μηχανισμοί από ότι πριν τη θέσπιση της υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης, πράγμα το οποίο δεν λέει και πολλά, για τους άλλους δεν δούλευαν πολύ καλά. Με πάση περιπτώσει, βασικό είναι ότι δεν λειτουργούν ικανοποιητικά, δεν προβάλλουν τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ενώσης και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό ουσιαστικά. Επίσης, στην παρουσίαση του δικτύου ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται μια παρατήρηση για μια ιστορική και εξωτερική σύνοχη, πράγμα το οποίο με βρίσκει ε, παρατήρηση που με βρίσκει σύμφωνο και δεν θέλω να τη συζητήσουμε και αργότερα. Έχω κάνει επίση δηλώσει στην Ολομέλεια που θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά. Έχουμε σημεία εστίαση, έχουμε την κατάρτιση και σε αυτά μπορεί να συμφωνούμε όλοι, αλλά πρέπει να περάσουμε και στην ουσία τη υπόθεση. Ε, είναι μια δουλειά που συνεχίζεται διαρκώς, είναι μια, ένα σεσίφιο έργο και βλέπουμε ότι μόλις τελειώνουμε ε, σε έναν τομέα πρέπει αμέσως να αρχίσουμε τη δουλειά κάπου αλλού. Ε, πρέπει όμως να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Επίσης, ως προς την υποχρέωση λογοδοσίας βλέπω κάποια κενά και στην έκθεσή μου θα τα συμπεριλάβω θα τα επισημάνω και ιδιαίτερα υπογραμμίζω το σημαντικό ρόλο που έχει διδραματίσει το Κοινοβούλιο ως προς τη διαφάνεια των επιδόσεων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στα θέματα της ε, συνεργασίας αυτής και νομίζω ότι μπορούμε πολλά πράγματα να επιτύχουμε εάν συνεργαστούν ε, η υποεπιτροπή μας με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και εν πάση πιστεύω ότι πολλά πράγματα πρέπει να καθίσανται γνωστά στην κοινή γνώμη, να βγαίνουν προς τα έξω για να υπάρχει αυτή η λογοδοσία. Δεν έχουμε αρκετή λογοδοσία. Δεν θα έχουμε ποτέ αρκετή λογοδοσία και αυτή είναι και μια από τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωση που πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Το γράφω αυτό Εσκεμένα λοιπόν στο κείμενό μου. Δεν διεκδικώ εκ μέρους του Κοινοβουλίου περισσότερες εξουσίες, αλλά απαιτώ να έχουμε περισσότερη λογοδοσία, διαφάνεια. Αφού μας λείπει. Επίσης δεν υπάρχει το στοιχείο της ισότητας. Ξέρω βέβαια ότι αυτό δεν ήταν προτίμηση της Δίας Άστον, αλλά πάντως δεν υπάρχει αυτό που θα έπρεπε να έχει ε, ιδιαίτερα υπογραμμιστεί και αντιμετωπιστεί, δηλαδή η ισότητα. Και κάτι ακόμη που ίσως κάποιοι μου πούν ότι δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα το υπογραμμίσω, πρόκειται για ένα ζήτημα κουλτούρας και νοοτροπίας, οργανωτικής δηλαδή κουλτούρας, την οποία θα χρειαστεί καιρό για να εισαγάγετε στην υπηρεσία σας και ξέρω ότι αγωνίζεστε να το καταφέρετε και σε από πλευρά σας. Ένας όμως από τους λόγους για τους οποίους δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί στα ανθρώπινα δικαιώματα εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο θα θέλαμε είναι ότι δεν έχουμε επαρκή γνώση και συνείδηση τη κουλτούρα των ανθρωπινών δικαιωμάτων σε επίπεδο ευρωπαϊκών υπηρεσιών εν γέννη. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει. Πρέπει να ενσπαρεί αυτή η ε, κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε και στη στρατηγική ε, αντίληψη στο, στρατηγικό σχεδιασμό που χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Χάου και την κυρία Γκόμεση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και θα ήθελα πρώτα να πω ότι συμφωνώ με τις δηλώσεις που ακούστηκαν μόλις τώρα από τον Ρούι Ταβάρες και από τον ε, κύριο Χόουιτ. Και θα συμπληρώσω ότι δεν υπάρχει τομέα στον οποίο να πρέπει να καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η νοοτροπία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, και να γίνει προσπάθεια της ενσωμάτωσης έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε συνέπεια, συνεκτική δηλαδή διαχείριση και χάραξη πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρωπινά δικαιώματα όπως ακριβώς υπογραμμίζει και η Διεθνής Αμνηστία όσο στον τομέα της ανάπτυξης. Τον τομέα ο οποίος καλύπτεται από τις αρμοδιότητες της, ε, του Επιτρόπου του Αρμόδιου για την Ανάπτυξη και που έχει να κάνει με χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερους δεσμούς. Παλαιούς δεσμούς σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή απεικιοκρατικούς, πράγμα το οποίο εξηγεί και την ιδιαίτερη εταιρική σχέση και στο πλαίσιο του Κοτονού. Απαιτεί επίσης εξάπαντος Ω αιχμή του δόρατο να προβληθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα το οποίο δεν διαπιστώνεται. Το άρθρο 896 ε, των, ε, της Συμφωνίας του Κοτονού και όλα αυτά τα προβλέπουν, αλλά αλλά όταν υπάρχει ένα σημαντικό χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο καλείται να ικανοποιήσει τον στόχο της ε, εκπλήρωσης των στόχων της χιλιετίας και ιδιαίτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα τα δικαιώματα της γυναίκας επισκιάζεται πολύ συχνά από το business as usual, της, ε, δηλαδή τρέχοντες, τρέχουσες εργασίες ε, και ιδιαίτερα τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Το Ταμείο Ανα... Ανάπτυξης όμως είναι το μόνο το οποίο δεν ελέγχεται από το Κοινοβούλιο γιατί δεν εγγράφεται στον προπολογισμό. Και ακριβώς αυτό το γεγονός εξυπηρετεί την αδιαφάνεια. Αυτό πρέπει να απαιτήσουμε λοιπόν. Πρέπει το Ταμείο Ανάπτυξης να εγγραφεί, να αρχίσει να εγγράφεται στον προϋπολογισμό, ώστε να υπάρχει και η λογοδοσία και η ε, διερεύνηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά όπως είπα χρειάζεται να ενσπαρεί αυτή η κουλτούρα των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Εδώ στις Βρυξέλλες, στις αντιπροσωπείες πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, υλοποιούμε τη Συμφωνία Κοτονού και τις λοιπές δεσμευτικές συμφωνίες που υποτίθεται πως προάγουν την ανάπτυξη. Αλλά χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει. Ευχαριστώ Άννα. Και η παρέμβασή σου μου θύμισε αυτό το οποίο έμαθα χτες σε μια συνεδρίαση της ε, εξωτερικής υπηρεσίας όπου γινόταν μια αξιολόγηση κάποιων μέσων και αυτό το οποίο έμαθα μεταξύ των οποίων του Ευρωπαϊκού Μέσου για Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πως ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη και η νοοτροπία και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όσοι παρακολουθούν αυτό το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ε, την επόμενη εβδομάδα στο Τρασβέργο παρουσιάζουν αυτή τη συνάδελφη και θα μπορούσαν να πάνε κάποια μέλη νομίζω του προσωπικού γιατί μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα ε, και νομίζω αυτό θα γίνει και στις 16 ε, Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες ε, και θα αφορά και την Επιτροπή μας. Οπότε νομίζω πως υπάρχουν πάρα πολύ καλές συστάσεις εκεί πέρα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα, κύριο κύριος Κούκαν. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στην ετήσια έκθεση «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο 2009» και την Ευρωπαϊκή πολιτική για το θέμα. Εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητάμε από την ε, ύπατη εκπρόσωπο να ξαναδεί ε, επανεξετάσει εκβάθρον την αποτελεσματικότητα όλων των ευρωπαϊκών ε, μέσων για τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις κατευθυντήριες γραμμές και για το Ευρωπαϊκό Μέσο για Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της διμερούς βοήθειας και της δράσης Ένωσης σε πολυμελή φόρα. Καλώς όριζω λοιπόν αυτή την κοινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την εξωτερική πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, δημοκρατία. Θα μπορούσε έτσι να υπάρξει μια ανακατάταξη των υφιστάμενων μέσων και των νέων μέσων για αποτελεσματικότερη προστασία και ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πολιτική μας. Η ανακοίνωση αυτή προτείνει δράση σε τέσσερις τομείς. Ε, τους νομικούς ε, μηχανισμούς, ε, ενσωμάτωση των πολιτικών, την ανάπτυξη σχέσεων και τον μία φωνή. Στόχο έχει να ενισχύσει την εμπλοκή της Ένωσης σε όλους τους τομείς ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτικά, ε, αστικά, οικονομικά και πολιτικά. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των μέσων και να επιφέρουμε ριζοσπαστικές αλλαγές για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους της συνθήκης της Λισαβόνας. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Παγκόσμια εμβέλεια φορέας θα πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο και βεβαίω φιλόδοξοι στόχοι απαιτούν φιλόδοξα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Η προσέγγιση της Ένωσης βεβαίως εξαρτάται από την κάθε χώρα. Δεν υπάρχει μία ενιαία μέθοδος, οπότε προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη και την πραγματικότητα έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα όπως αναφέρθηκε και στην παρέμβαση του κυρίου Ποπόφσκη. Η ύπατη εκπρόσωπος έχει δεσμευτεί να ασχοληθεί με συγκεκριμένα οριζόντια θέματα για τα επόμενα τρία έτη. Την δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να ενσωματώσει ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις πολιτικές δηλαδή ανάπτυξιακή συνεργασία, εμπόριο, αντιτρομοκρατία, διαχείριση κρίσεων, πρόληψη συγκρούσεων και διακυβέρνηση του διαδικτύου. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια μέσα ε, με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να να αναλάβει ένα ισχυρότερο ρόλο. Actions and participation in the EU. Πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα του ΟΗΟ στην τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΑΣΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμούς. Και να βρεθεί ένας τρόπος να ακουστεί καλύτερα η φωνή της Ένωσης. Ενωμένοι βεβαίως είμαστε ισχυρότεροι και με το να μιλάμε με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δύναμη να προσφέρει θετικά στον κόσμο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Κομισιών και Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγγυηθεί πω το μήνυμά τη θα ακουστεί ε, άνα τον κόσμο με τρόπο συντονισμένο. Δυστυχώς ε, αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν π.χ. όσον αφορά την ε, τοποθέτησή μας στον ΟΗΕ. Πρέπει να σκεφτούμε την ε, αποτελεσματικότητα διαλόγου με χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία είναι προφανές πως ε, ο διάλογος δεν έχει κανένα νόημα στις χώρες εκείνες όπου δεν παίρνουν σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν υπάρχουν αυτά αποτελέσματα. Επίσης οι ρήτρε στις συμφωνίες με τρίτες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου συχνά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, αλλά η αποτελεσματικότητα των ρητρών αυτών βεβαίως εξαρτάται και από τη δυνατότητα επιβολής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην 19η συνεδρίασή του θα εξετάσει την συνενοχή ευρωπαϊκών εταιριών στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της Ένωσης. Καλούμε λοιπόν την Βαρόνια στον να εργαστεί σε κατεύθυνση σύσταση ενός συστήματος κυρώσεων για να παρακολουθεί τέτοιες περιπτώσεις και να φροντίσει οι εταιρείε αυτές να μην λαμβάνουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ή οποιαδήποτε βοήθεια από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η κοινή ανακοίνωση που συζητήσαμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα προτείνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια πράγματα για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων αυτών. Οπότε βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρει στη διαδικασία αυτή. Και, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να ομολογήσουμε πως αν ήταν ε, εδώ η κυρία Αντρικιένε, τα ίδια ακριβώς θα έλεγε ε, που είπα και εγώ. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Kukan, for your very... Ευχαριστώ κύριε Κουκάν. Πληρέστατη παρουσία σας. Με ιδιαίτερη προσοχή άλλωστε. Άκουσα και εσάς και την κυρία Αντρικέινα. Και ο κύριος Χάουτ και ο κύριος Ταβάρης και εσείς υποστηρίξατε αυτές τις ιδέες. Τη μεταρρύθμιση του δικαστικού, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν γυναίκες και παιδιά ιδιαίτερα σε κατάσταση ε, εμπόλεμη, την προστασία μάλλον των παιδιών και των γυναικών απογραμμίζουμε ιδιαίτερα ότι είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στις ευθύνε ε, του επιχειρηματικού κόσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις λοιπές χώρες. Και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ποπόφσκι, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. μίλησε για τη συνεδρία συγκέμνηχε ο κύριος ε, Παπόφσκι στις αρχές Μαρτίου στην Κοπενχάγη με τις ε, ε κυβερνήσεις. Και ο Δανός υπουργό όταν μίλησε στην ΑΦΕΤ υπεγράμμισε ότι οι Γερμανοί δηλαδή η δική μου κυβέρνηση έχουν αποστείλει μία επιστολή για την αναθεώρηση και άρα υπάρχει σχετική παρακολούθηση αυτό όμως δεν αρκεί. Γι' αυτό παρακαλώ όσοι έχετε πρόσβαση στις κυβερνήσεις σας, επιμείνετε. Έρθετε σε επαφή μαζί τους. Να μην μιλάνε μόνο, να μην περιορίζονται μόνο στα λόγια, αλλά να τα μετατρέπουν και σε έργα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους υπουργούς τις ευθύνες τους. Έχουμε επίσης τι ε, κυβερνήσεις και εμείς, αλλά θα πρέπει να, το να επιμείνουμε. Επίσης, πρόταση, ε, έκθεση καλύτερα γενικότερη του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση αυτή για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης ε, και εξέταση του τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να βελτιωθεί που θα μας ε, καθιστούσε πολύ πιο ευχερή την υλοποίηση αυτή, την παρακολούθηση μάλλον της υλοποίησης αυτής θα πρέπει να αναπτυχθεί. Ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο σχέδιο, αλλά δεν πρέπει να το ε, αμελήσουμε. Πρόκειται για μια πολύ καλή ευκαιρία. Και πρέπει να απευθύνουμε έκκληση και στα άλλα όργανα να πάρουν πιο πολύ στα σοβαρά την υπόθεση αυτή. Αν μπορούμε να το καταφέρουμε για, για την ανάπτυξη, ασφαλώς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τότε λοιπόν μπορούμε για το πρόγραμμα δράσης και την ουσιαστική αναθεώρηση να ξεκινήσουμε εκ παραλίλου με τη θέσπιση ενός, μιας ομάδας συντακτικής από τα θεσμικά όργανα που θα επεξεργαστεί μια κοινή διακήρυξη. Πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει σχετικά ευχερός θα υποβάλω τη σχετική σύσταση. Ο κύριος Ποπόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Μας ενθαρρύνεται να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για να απαντήσουμε στα όσα ακούστηκαν. ζήτημα κουλτούρας που ακούστηκε ότι λείπει. Πρέπει λοιπόν ε, να συζητήσουμε και τα χρονοδιαγράμματα και τον ορισμό βεβαίως του, του εκπροσώπου. Ε, αλλά πέραν αυτού, αλλαγή, ε, η πρόκληση, συνοχή το έργο αυτό της υλοποίησης θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Επιτροπή σε διάφορους τομείς, όπως το εμπόριο, Φερρυπίν. Η μετανάστευση και άλλες τομεακές πολιτικές ώστε να επηρεάσουμε ή να ευαισθητοποιήσουμε το ΣΥΠΗΝ άλλες πολιτικές σε τέτοια σημαντικά θέματα. Δυνατότητα θα μπορούσαμε να είχαμε χάρη στο πρόγραμμα ή στα μέσα, τα εξωτερικά μέσα για το, μέσα στο πολιετές οικονομικό πλαίσιο που θα έχουμε, όπου συμμετέχει το Κοινοβούλιο για τις συναποφασίση για τον εαυτό σύνολο όμως ε, οριστικοποιούνται ταυτόχρονα και οι κατευθύνες γραμμές. Και θα πρέπει θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διακυβέρνηση, ζητήματα δηλαδή τέτοια, να εξετάζονται ευρύτερα και όχι μόνο άπαξ και προγραμματιστεί το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Δημοκρατία και τα Ανθρωπίνα Δικαιώματα. Σε ευρύτερο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην αναπτυξιακή πολιτική Φερρυπίνη, στο σχετικό μέσο ή και στο αναπτυξιακό ταμείο. Θα πρέπει ήδη να περιλαμβάνονται αυτά και αποτελεί αυτό μια καλή ευκαιρία, πιστεύω, ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να λαμβάνονται υπόψη. Θα επανέλθω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη λίγο. Πάντως, ε, θα ήθελα να πω ότι ήδη έχουμε ένα δίκτυο αντιστοίχηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων σε όλες τις αντιπροσωπείες βεβαίως ή μάλλον α, α, αντεπιστελόντων μελών στις αντιπροσωπίες βέβαια δεν έχουμε πάντα τόσο πολύ προσωπικό και χρόνο αλλά υπάρχει ένα δίκτυο και άρα αποτελεί αυτό μια καλή βάση ταυτόχρονα στις αντιπροσωπείες αλλά και στα κεντρικά γραφεία έχουμε επικοινωνία με τρεις συγκεκριμένε και εξειδικευμένες συνεδριάσεις κάθε χρόνο και θα σπίσουμε ταυτόχρονα ένα δίκτυο των ε, σημείων εστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις, ε, με, με όρους γεωγραφικούς πλέον της επίδεσης εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό συνεχίζεται. Θα χρειαστεί χρόνος για να αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα που αναφέρατε, αλλά πρόοδο σημειώνουμε. Και ελπίζω ότι θα καταστεί και πιο ορατή για σας, για τις υπηρεσίες μας, την προσωπή μας, τα επιτοπογραφεία μας, σύντομα. Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη. Βεβαίω πρόκειται για ζήτημα συνοχής, αλλά επίσης και όπως ανέφερε η κυρία Γκόμες, Όταν εξετάζουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για, την, ε, για το μέλλον της πολιτικής ανάπτυξης, Agenda for Change όπως ονομάζεται, βλέπουμε ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και άρα αυτό πιστεύω θα αποτελέσει τον μύτο της Αριάδνης για τα επόμενα χρόνια. Και θα επηρεάσει τον τρόπο λειτουργία των χρηματοπιστωτικών μέσων. Επίση όταν μιλάμε για το μέλλον, υποστήριξη δημοσιονομική προς, του τους θα πρέπει το στοιχείο αυτό να υπογραμμιστεί ιδιαίτερο. Τα ανθρωπινά δικαιώματα δηλαδή και η δημοκρατία. Ε, παραδείγματι, προτείνουμε συμβάσεις διακυβέρνησης τους εταίρους, που θα ήταν κάποια συμβόλαια που θα δεσμεύουν του εταίρου σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Βεβαίω αυτό θα πρέπει να το συμφωνήσουν και τα κράτη-μέλη. Αποτελεί όμω μια ιδέα που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο, μια προσέγγιση που θα διεκδικούμε όλο και περισσότερα, όπως ε, λίγο πολύ έχουμε δει και στην ε, πολιτική γειτονία, όπου θέλουμε περισσότερη, καλύτερη διακυβέρνηση, ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να, και να τους πει στρίξουμε σε αυτό το έργο. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Τα μέσα που αναφέρθηκαν Φιρπίν, ε, διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διακυβέρνηση υπό το 96 άρθρο της ε, Συμφωνίας του Κοτονού. Για το χρονοδιάγραμμα, το αναφέρατε κι εσείς, μέχρι τον Ιούνιο. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε κατά πόσο συμπίπτει με την εργασία σας, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε διευκρίνηση ως προς τον ε, ε, διορισμό του ειδικού συμβούλου δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ε, περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο, οπότε θα έχουμε και ένα πρόγραμμα δράσης από το Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει αυτό το νέο πρόσωπο να συνεισφέρει στην εφαρμογή του έργου μας. Δεν μπορώ να πω κατά πόσο θα γίνει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Θα πρέπει να ορίσουμε επακριβώς την εντολή και η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της ΥΠΑ εκπροσώπου. Αλλά πρόθεσή της είναι να μην ε, περιμένουμε πολύ, γιατί αυτό θα προωθήσει και τον ορίζοντα της κοινή μα εργασίας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάτι τέτοιο συμβαδίζει και με την δήλωση περί της ΥΠΑ της εκπροσώπου γιατί α, ακριβώς θα ήθελε να μιλήσει και για θέματα λογοδοσίας πριν ο η υπεύθυνη αναλάβει τις εργασίες της. Εν συμπεράσματι, ευχαριστώ πολύ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Θα σας ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη συνεχιζόμενη εργασία Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να είμαστε πειθαρχημένοι και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Κύριε Ποπόφσκι, θίξατε στο τέλος ένα θέμα για τον διορισμό ε, ενός ή μίας εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για μας ε, στην Επιτροπή μας, στην Υποεπιτροπή μας. Θα θέλαμε να ακούσουμε αυτό το πρόσωπο, όπως γίνεται και σε επίπεδο ε, ΑΦΕΤ. Δηλαδή, όχι να μας, ε, να μας παρουσιάσετε απλώς τον, την διορισμένη, αλλά να γίνει μια σαν μικρή ακρόαση πριν. Υποθέτω, λοιπόν, ότι οι πολιτικές ομάδες θα δουν, θα ορίσουν τους σκιώδεις εάν δεν έχει ε, προαποφασιστεί και θα μπορέσουμε να αρχίσουμε με τις εργασίες μας. Τώρα φτάνουμε στο επόμενο σημείο που είναι η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μιλώντας και για την στρατηγική πολιτική στον τομέα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συγκεκριτή είναι ο Ρίτσαρντ Χάουιτ. Έχουμε και τους ε, σκιώδεις Ντόνσκι από το Άλτε, Βερζιά από την Γκουέ και Τάνοκ από τους Ευρωπαίους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Επίσης, τον κύριο Ταβάρες από τους ε, ε, πρασίνους. Έχουμε και τον ε, κύριο Σουάν από την ΕΙΕΔ, ο οποίος θα μας απαντήσει. Έτσι βλέπω από τις σημειώσεις μου. Και δεν θα ήθελα να πω πολλά εκ των προτέρων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χάουιτ, στον εισηγητή. Και να πω ότι η έκθεση σας έχει δοθεί σε όλες τις γλώσσες. Κύριε Χάουιτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας, όπως και πριν, πως υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία και πολλές καθυστερήσεις και πολύ σημαντικά ζητήματα σύνοχης για διάφορες εκθέσεις πολλών εισηγητών και είναι σημαντικό η έκθεση αυτή να μην αλλάξει κάποια πράγματα που αναπτύξαμε αλλά να τα ενισχύσει. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνεργασία και ελπίζω να το δούμε αυτό στο σχέδιο κειμένου, ειδικά στη στρατηγική αναθεώρηση. Οπωσδήποτε είναι δύσκολο ε, αυτό το κομμάτι να συνταχθεί, αλλά προσπάθησα να μείνω στο πνεύμα της συμφωνίας. Υπάρχουν αρκετά σημεία που λένε πως θα υπάρξει μία λεπτομερής έκθεση και βεβαίω ε, θα δούμε και τις λεπτομέρειες ε, εκεί πέρα και βεβαίω θα συνεργαστώ με τους και και είμαι βέβαιος πως θα συμβεί αυτό. Επίσης, νομίζω πως η συζήτηση τωρινή για το Ταμείο περί Δημοκρατίας είναι θετική. Δεν χρειάζεται νομίζω να τσακωθούμε γι' αυτό. Και γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση αυτή τη στιγμή για το πώς θα προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Και αυτό το οποίο θα έλεγα επίσης ε, επί της διαδικασίας νομίζω πως μπορούμε να πούμε στους συναδέλφους της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης πως φέτος δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ το Κοινοβούλιο με την ετήσια έκθεση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και νομίζω πως η συνεργασία με το Κοινοβούλιο έπεσε θύμα των διαδικαστικών ε, δυσκολιών. Δεν ξέρω αν ήταν εσκεμμένο Ξέρω πως η γραμματεία μας έστειλε πληροφορίες, δεν το αμφισβητώ, αλλά η ετήσια έκθεση θα πρέπει να είναι η ετήσια έκθεση της Ένωσης και όλων των θεσμικών οργάνων και θέλουμε η γραμματεία μας να εμπλακεί πλήρως στην σύνταξη αυτής και ελπίζω να γίνει αυτό τα επόμενα χρόνια. Αυτά για τα διαδικαστικά. Επειδή είναι λοιπόν συνολική αυτή η ετήσια έκθεση, υπάρχουν πολλά πράγματα, δεν θα τα σχολιάσω όλα. Βεβαίω θέλω να ακούσω τι θα πούν οι σκιώδεις αν θέλουν, αν έχω κάνει κάποιο λάθος, αν έχω παραλείψει κάτι. Θέλω να ακούσω λοιπόν από τους συναδέλφους τι θα γίνει και δεν μπορώ βεβαίω να καλύψω τα πάντα. Αλλιώ οπωσδήποτε θα τελειώσει ο χρόνος. ειδικά σε σχέση με το ότι οι εκθέσει εκθέσεις ε, ε, είναι πολύ περιγραφικές αλλά δεν προτείνουν καμία δράση. Και αυτό οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει. Και το ζήτημα της ενσωμάτωσης πολιτικής, τα είπε και ο κύριος Ποπόφσκι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δεν ακούγεται έτσι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό. Να περάσω λοιπόν απευθείας στην παρουσίασή μου για τους νέους τομείς που προσπαθούμε να θίξουμε φέτος ζητήματα πολύ σημαντικά όχι μόνο η Αραβική Άνοιξη αλλά η εξέγερση στη Βυρμανία οι αποτυχημένες νομίζω μπορούμε να πούμε εκλογές στο Ιράν που έθεσαν ζητήματα δημοκρατικής μετάβασης και αυτό το οποίο η Βαρόνι Άστον λέει βαθιά δημοκρατία, όχι μόνο δηλαδή ε, δίκαιες εκλογές, αλλά το τι προηγείται και το τι ακολουθεί. Είδαμε λοιπόν πραγματική πρόοδο προς την κατάργηση της ανατικής ποινής, πρέπει να το πούμε αυτό. Είδαμε επίσης την δέκατη επέτειο του ψηφίσματος Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες ε, και την ασφάλεια το 1325 για να εξετάσουμε το ρόλο των γυναικών στην ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το αναφέρουμε στην έκθεσή μας και βεβαίως ε, είδαμε τα συμπεράσματα της εξέτασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω καλά τα πήγε στο να στηρίξει εντολές για ειδικού απεσταλμένους ε, και βεβαίως δεν τα καταφέραμε όλα όσα θέλαμε στον ΟΗΕ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν τα πήγε καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το αναγνωρίζουμε αυτό στην έκθεσή μας. έτσι φέτος είδαμε και το λέω σαφώς στο κείμενο, μια καθυστέρηση σε σχέση με την κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ΕΣΔΑ και επίσης υπήρχαν ανησυχίες για αντιτρομοκρατικούς νόμους και στις δικές μας χώρες και σε τρίτες χώρες και για το πόσο συμβιβάζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το βάζω στο σχέδιο παρά το ότι βεβαίως είναι ευαίσθητο ζήτημα και οπωσδήποτε ε, και εγώ δεν είμαι υπέρ των τρομοκρατών, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να σεβαστούμε το, το κράτος δικαίου, γιατί αυτό ακριβώς θέλουν να υπονομεύσουν. Υπάρχουν επίσης νέες ιδέες στο κείμενο. Ε, θα αναφέρω κάποιες για να υπάρξει ενδιαφέρον. Θέλω να δω αν τις υποστηρίζουν οι συνάδελφοι. Αναφέρω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Νίκολς περί ενός μηχανισμού εσωτερικής και εξωτερικής συνέπειας πως δεν υπάρχει δηλαδή ένας τέτοιος μηχανισμός και επίσης για ζητήματα σύλλου και μετανάστευσης ε, για την ομάδα εργασίας δεν είναι αυτό η απάντηση στο πρόβλημα αλλά είναι μια προσέγγιση και το βάζω αυτό στην έκθεση επίσης ε, επί σειρά ετών λέμε πως πρέπει να υπάρχουν δείκτες μετρήσιμοι της προόδου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ειδικά στο πλαίσιο της πολιτικής περισσότερα για περισσότερα της Βαρόνης Άστον που πρέπει να μεταφραστεί κάποτε και σε λιγότερα για λιγότερα γιατί το να διακόπτουμε τις εμπορικές σχέσεις με κυρώσεις είναι ένα πολύ έτσι, άμβλη μέσο πρέπει να δούμε επίσης το πόσο θα γίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα τμήμα των εμπορικών συμφωνιών. Λέμε επίσης ε, πως η κύρωση των διαταξιών της ε, Ρώμης θα πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για εμπορικές παραχωρήσεις και του γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων καθώς επίσης και η υπογραφή του πρωτοκόλλου περί βασανιστήριων και βεβαίως ενσωμάτωση της πολιτικής αυτής όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο τι κάνουμε στον ΟΗΕ. Ενσωμάτωση με το να δούμε τις συστάσεις άνα χώρα και να τις βάλουμε στην στρατηγική της κάθε χώρας, στο, τα θέτουμε στο διάλογο που έχουμε με την κάθε χώρα να λέμε ε, να πούμε επίσης πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον προπολογισμό του Διεθνούς ε, Ποινικού Δικαστηρίου αυτό το έχουμε πει από την έκθεση Chrysler Φλερίδη και το αναφέρω όπως είπα και πριν πως ε, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι δεν λειτουργούν και παρά τα επίσημα αιτήματα του Κοινοβουλίου η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν μου έδωσε την αξιολόγησή της για τον διάλογο με την Κίνα. Νομίζω πως και πως το παρελθόν ε, μας είχε επιτραπεί να πάμε σε, μια, σε ένα σκοτεινό υπόγειο ε, της Κομισιόν και να διαβάσει αλλά δεν είναι καταστάσεις αυτές τώρα, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι αυτή η απέτηση, ε, δεν πληρώνεται έτσι η απέτηση που υπάρχει για ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Πρέπει να αλλάξει αυτό άμεσα και απαιτώ πρόσβαση σε αυτές τις αξιολογήσεις. Για το θέμα, ε, θέσαμε και το θέμα των λευκών γάμων, των ψεύτικων με συγχωρείτε, των α, καταναγκαστικών γάμων. είναι αδιανόητο το ότι δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Επίσης, Θα ήθελα ε, και τροπολογίες από τους ε, συναδέλφους για το θέμα αυτό και τα διεθνή μήμια. Θα με ενδιαφέραν κάποιες ιδέες λοιπόν και να πω στην πράσινη ομάδα ως εισηγητής του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Εμείς πρέπει να χρησιμοποιούμε την ε, ορολογία ε, επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί κοιτάξτε, ε, πολλά πράγματα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μη δεσμευτικά. Εμείς πρέπει να πούμε πως είναι καθήκον των επιχειρήσεων να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να χρησιμοποιούμε την, ε, τη σωστή ορολογία και όχι την ορολογία εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αλλιώς υπονομεύουμε αυτούς και αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Κούκαν είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά αυτή η μελέτη του Εδιμβούργου, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια όσον αφορά μελλοντικέ δράσεις και την αναφέρω στο κείμενό μου και Νομίζω πως υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να το κάνουμε αυτό λοιπόν, νομίζω θα πάμε καλά στο μέλλον. Θα κάνουμε και εμείς μια ακρόαση βεβαίως στην υποεπιτροπή μας, την οποία αναμένω. Αρκετά πράγματα λοιπόν περιέχονται, ελπίζω να τα ανέφερα όλα και αναμένω τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και ελπίζω να διαμορφώσουμε μαζί το κείμενο για να έχουμε ένα όσο το πιο φάρο ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω λόγο στους Κιώδης. Ποιος θα ήθελε το λόγο? Ο κύριος Σίπ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι αυτό το σχέδιο έκθεσης μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλά συγκροτημένο σε παρόμοια έγγραφα τα οποία έχουν τόσο ευρύ περιεχόμενο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και δεν μιλώ μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώ για ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να δεχτεί και άλλες ε, υποδείξεις. Θα μπορούσαμε να εντάξουμε και άλλες υποδείξεις σε αυτή την ε, έκθεση. Νομίζω όμως ότι η εργασία και οι τροπολογίες μας θα βοηθήσουν έτσι ώστε να φτάσουμε σε έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ Χάουιτ και Σκιωδών. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε πολύ καλά. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή σε ένα σημείο. Νομίζω ότι θα ήταν ε, σκόπιμο να αναφερθούμε στη δήλωση της Κορεπέρ της 15ης Δεκεμβρίου. Ο κύριος Χαουίτ υπέβαλε προτάσεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και μια αναφορά στην Κόρεπερ, στις δηλώσεις της Κορεπέρ. και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 1 η Δεκεμβρίου που έθιξε και το θέμα της πολιτικής γειτονίας και τα συμπεράσματά μας μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα στα πλαίσια της Αραβικής Άνοιξης πολλά ελέγχθησαν καθώς και για την πολιτική γειτονία. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα χωριστά. Και υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις της Αραβικής Άνοιξης. Πιστεύω ότι στην έκθεση Βερονίκ Κάιζερ αυτό το θέμα ήταν ένα από τα πρωταρχικά θέματα, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα ειδικό Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση Εδώ γίνεται λόγος μόνο για την ε, ε, πρωτοβουλία αυτή, χωρίς να επεκταθούμε. Επίσης κάτι άλλο. Στο σημείο 64 μιλάμε για την ε, Διεθνή Κατάταξη Ασθενειών. Νομίζω ότι σε χώρες όπως η δική μου θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις υποδείξεις των πολιτικών και να μιλάμε για μια γενικότερη κατάταξη. Νομίζετε όμως ότι είναι απολύτως αναγκαίο. Γιατί ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση στο πρώην κομμουνιστικό μπλοκ, Ρουμανία, Κίνα, Κούβα εδώ είχαμε ε, ειδικέ εκθέσεις που αφορούσαν το θέμα της σχιζοφρένειας. Και η σχιζοφρένεια ήταν μια ασθένεια η οποία κατατασσόταν ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πού γίνονται πολιτικές διώξεις και πώς μπορούμε να κατατάξουμε ορισμένες ασθένειες ή να δούμε κατά πόσο ε, κατατάσσονται σωστά. Στην ετήσια αυτή έκθεση νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για την ποιότητα αυτού του εγγράφου και είπαν ότι θα πρέπει να μην επαναλαμβάνουμε αυτά που είχαμε πει τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει δηλαδή να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα θέματα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για το μέλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς μιλάτε για το ότι αυτή η έκθεση μιλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και το πώς θα κινηθούμε γενικότερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ειδικά θέματα. Δεύτερον, υπάρχει μία σειρά εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως και θα πρέπει να το δούμε αυτό και μέσα στα πλαίσια των εξαμήνων. Υπάρχουν εκθέσεις του Human Rights Watch, του Freedom House, που θα πρέπει να δούμε πώς θα τις εντάξουμε. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία μας όταν θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τελική μορφή στη δική μας έκθεση. Θα πρέπει να γίνει μνήα και σε αυτές τις εκθέσεις για να βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. γιατί από αυτές τις εκθέσεις έχουμε πληροφορίες από άλλες πηγές για να δούμε πώς γίνονται αξιολογήσεις ως προς ειδικά θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο βασιζόμαστε στις γνώμες, στη γνώμη των συντακτών αποκλειστικά ή αν υπάρχουν άλλες πηγές. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις πηγές. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Κάτι άλλο τώρα. Ένα βασικό θέμα, ένα θέμα που με απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα στην έκθεση αυτή να γίνει μία στις εθνικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί διαδραματίζουν όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες όπου υπάρχουν και προτιμησιακές σχέσεις. Δηλαδή ε, χώρες όπου αναπτύσσουμε σχέσεις γειτονίας προς Ανατολάς. Να δούμε ε, δηλαδή πώς προωθούν ε, αυτά τα θέματα οι εθνικές οργανώσεις. Η συνήγορος του πολίτη στην Πολωνία έχει προωθήσει τέτοια θέματα και πιστεύω ότι τη στιγμή που μιλάμε για νέα δημοκρατικά συστήματα περνώντας από απολυταρχικά στο νότο της Μεσογείου θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα σημασία Θα πρέπει να δούμε επίσης πώς κινείται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα εγκλήματα σε διεθνές επίπεδο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν γίνεται μνήα για τα θύματα. Τι γίνεται για την αποκατάσταση τους, για την αποζημίωσή τους. Το θέμα των θυμάτων είναι ύψης της σημασίας, κύριε Χάουιτ και θα πρέπει να το δούμε και μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Νομίζω ότι εάν λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στο ε, Σύμφωνο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα πρέπει να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήρθαμε σε επαφή και με τον ε, συνήγορο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα πρέπει να το δούμε ως θέμα μεταξύ ομοτήμων και όλα αυτά να ενταχθούν και στην έκθεσή σας, ε, κύριε Χάουιτ. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα διάφορα ε, σχέδια και προγράμματα μεταξύ ομοτήμων μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να προωθήσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Μέσο για τις πρωτοβουλίες αυτές για τη συνεργασία των ε, συνηγόρων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ανατολικής Ευρώπης. Ε, τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για το εξής. Θα πρέπει να υπάρξουν ε, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του βραβείου Ζαχάροφ έχουμε προβεί στη σύσταση ενός δικτύου των βραβευθέντων έτσι ώστε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν στη Βυρμανία. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε το θέμα, τα θέματα των βραβευθέντων Συμφωνώ με τον κύριο Χάουιτ ότι θα πρέπει τα θέματα αυτά να προωθηθούν ως προς τα δίκτυα πληροφόρησης, διότι βλέπουμε κάτι το εξαιρετικό ως προς την επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Το βλέπουμε και στην κύρωση της άκτα βλέπουμε ότι δεν ε, υπερασπιζόμαστε επαρκώς το θέμα του ιδιωτικού βίου. Θα πρέπει να το προωθήσουμε και στην Πολωνία και αλλού. Τελευταία παρατήρηση. Το θέμα των θρησκευτικών διώξεων. Βλέπω ότι το θέμα προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Πολλές φορές διώκονται ε, πρόσωπα για τον θρησκευτικό τους προσανατολισμό. Το βλέπουμε στις, ε, στους διωγμούς των χριστιανών παγκόσμια και ιδιαίτερα στη Βόρειο Κορέα, αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Βλέπουμε ότι προωθούνται αυτές οι διώξεις και στο Ιράκ και στην Αίγυπτο. Βλέπουμε τι γίνεται με τους κόπτες στην Αίγυπτο. Θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των διώξεων αυτών. Έχει μεγάλη σημασία η υπεράσπιση των μειονοτήτων, των θρησκευτικών μειονοτήτων. Θα πρέπει να το έχουμε κατά νου σε όλες μας τις διαπραγματεύσεις. Thank you. Ευχαριστούμε κύριε Ζήπ. Είμαι σίγουρη πως ο άκουσε τις συστάσεις σας. Τώρα έχουμε δύο ακόμα σκιώδεις εισηγητές. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ντόνσκι και μετά η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Χάουιτ και αυτό το οποίο είχε μεγάλη σημασία ήταν το ότι συμβουλευτήκαμε τους συναδέλφους μας και τις άλλες πολιτικές ομάδες, γιατί νομίζω πως κάθε συνάδελφος θεωρεί πως υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά την ετήσια έκθεση, γιατί μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ε, τα γεγονότα επιτόπου ή δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες όλων των χωρών. Γι' αυτό επιφελούμαστε κάθε φορά από αυτό το διάλογο πολιτικών ομάδων, συναδέλφων και νομίζω πως η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική από τη σκοπιά της αξιολόγησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τονίζει ο εισηγητής πως αντί για περιγραφή ανεξαρτήτως του πόσο καλή μπορεί να είναι αυτή η περιγραφή πρέπει να γίνεται και μία αξιολόγηση γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις. Η ετήσια έκθεση δεν ε, αντιμετωπίζει μόνο τις αδικίες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την αδιαφορία, που είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και δεν μιλάμε μόνο για την πολιτική ελίτ, αλλά ακόμη και το ότι η περιγραφή μπορεί να είναι πολύ λεπτομερής, αλλά εάν δεν έχει αξιολόγηση, εάν δεν έχει κάποια ηθική βάση, νομίζω πως δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο που προσφέρουμε στον κόσμο. Γι' αυτό νομίζω πως έχει μεγάλη σημασία η αξιολόγηση. Και συμφωνώ πλήρως. Ε, κάτι άλλο το οποίο κάνει ιδιαίτερη αυτή την έκθεση είναι πως γνωρίζουμε πως ένα πρόβλημα που είναι κοινό μυστικό μεταξύ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια επιλεκτική προσέγγιση. Ξέρουμε πως έχουν προτεραιότητες οι συνάδελφοί μας ε, ε, τις θρησκευτικέ ομάδες, άλλοι συνάδελφοι τους ε, ΛΟΑΤ και κάποια πράγματα ορισμένες φορές δεν μπορούμε να τα συζητάμε γιατί πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας και από αυτή την πλευρά της συνολικής έτσι, νομίζω πως αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα η έκθεση. Και η εντύπωση μου είναι πως μία από τις δυσκολίες που έχουμε τώρα ε, είναι πως αντί για τις πολύ προφανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως την εποχή του ψυχρού πολέμου τώρα αντιμετωπίζουμε το ότι κάποιες ε, παραβιάσεις είναι κάπως πιο δύσκολες το να διαπιστωθούν όταν μιλάμε για την ελευθερία στο διαδίκτυο ή το αν υπάρχει μια νοοτροπία παραδείγματο χάρη, η νοοτροπία της ατιμορρησίας των πολιτικών ή το ειδικό καθεστώς ε, των νομοθετικών οργάνων σε κάποιες χώρες. Νομίζω λοιπόν πως γίνονται πολύ πιο αφηρημένα τα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπειρογνώμονες, να έχουμε εμπειρικά δεδομένα και ταυτόχρονα να υπάρχει ένα πνεύμα συναδελφικό. Γενικά πρέπει να πω πως η έκθεση αυτή ωφέλησε, από πολλά διδάγματα θέλω και πάλι να εκφράσω την ευγνώμοσύνη του. Νομίζω πως εγώ τουλάχιστον επωφελήθηκα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντόνσκης. Καθώς συμφωνώ απολύτως ότι πάντα με πολύ μεγάλη χαρά συνεργαζόμαστε με τον κύριο Χαουίτ που δέχεται πάντα τη συμμετοχή μας και την Ουθαρίνη. Η δε προσέγγιση του πιστεύω εμπλουτίζει τον τακτικό ετήσιο κατάλογο και αποφεύγει και μια ε, προσέγγιση την οποία θα αποκαλούσα σχετική ρελατιβιστική. και μας επιτρέπει μια πιο γενική προσέγγιση με διαφορετικά πρίσματα σε μια χρονική στιγμή όπου όντως χρειάζεται περισσότερη συνοχή. για τις εκθέσεις και τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται αναδιοργάνωση βέβαια, αλλά και πέραν αυτού, περισσότερο από ό,τι ποτέ, συνοχή μεταξύ λόγων και έργων. Θα ήθελα λοιπόν, γιατί κάποιες παράγραφοι μου φαίνονται, φαίνεται ότι χρειάζονται συζήτηση, να συζητήσουμε λίγο την συνοχή εσωτερική και εξωτερική, θεωρώ πολύ σημαντική. Θα ήθελα επίσης να επικεντρωθούμε στα θέματα τα σχετικά με το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα. και κυβερνοεγκληματικότητα, καθώς και τους νέους τύπους δημοκρατίας, ε, η προσέγγιση δημοκρατίας που αναπτύσσονται ε, μέσα από το ίντερνετ. Πρέπει να επαγρυπνούμε ιδιαίτερως για να αποφύγουμε την απώλεια εστίασης και αλλαγή εστίασης σε σχέση με το επιδιωκόμενο και την ε, μετάβαση σε συστήματα πιο πολύ εστιασμένα στην ασφάλεια παρά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης θα ήθελα στο θέμα των ε, ασυνεπιών να αναφερθώ, γιατί ήταν ε, κάτι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα με εξόριξε πραγματικά. Μίλησε για συνοχή και συνέπεια ο κύριος Χάουιτ και επαγρύπνηση ως προς την αραβική άνοιξη. Συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε σε πολιτική επαγρύπνηση. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω το, ότι τα όσα πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο χώρο της εταιρικής σχέσης με την Ισία με εξοργίζει με κάνει ε, έξω φρενών και το λέω αυτό, θα περιγράψω πιο συγκεκριμένα, με δύο παραδείγματα. Τι εννοώ. Εκεί όπου λέγεται ότι θα πρέπει η ταχύτητα να θεσπιστεί η Επιτροπή Επιχειρηματιών, ε, την Ισίων ε, και Ευρωπαίων, αλλά τα ζητήματα των πολιτικών ελευθεριών τα αφήνουμε, τα παραπέμπουμε στις καλένδες μήνυμα κάκιστο για τέτοιες χώρες και επίσης ε, επιμένουμε στις ε, διάφορες πολιτικές για απελευθέρωση των αγορών, ελεύθερες συναλλαγές, ελεύθερες πολιτικές, πολύ περισσότερο από ό,τι στις ανάγκες οικονομικές και κοινωνικές της Τινησίας. Μπορεί να σας φαίνεται κάπως χονδροειδής η περιγραφή, αλλά ε, η συζήτηση για την βελτίωση του τουρισμού στην Τινησία, στην Επιτροπή, πέρασε μέσα από την απελευθέρωση των αερομεταφορών. Μα το πρόβλημα στον ε, τουρισμό της Τινησίας δεν έχει να κάνει ούτε με τον ανταγωνισμό, ούτε με, τις, ε, με την ανυπαρξία ενδεχομένω ε, παρκών μέσων. Τον αντίον μάλιστα οι τιμές τουλάχιστον είναι από τις πιο χαμηλές για την Τινησία αεροπορικές μεταφορές. άρα λοιπόν δίνουμε εσφαλμένα μηνύματα. Είναι καταστροφική μια τέτοια δράση. Η Τινησία είναι άλλωστε η χώρα εκείνη η οποία είναι περισσότερο σε θέση να προχωρήσει από τις άλλες αραβικές χώρες και άρα μπορούμε να έχουμε ένα πρίσμα ε, μέσα από το οποίο θα μπορούμε να εξετάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα μετά την Αραβική Άνοιξη και τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ε, οικουμενικών ανθρωπινών δικαιωμάτων που δεν μπορούμε βέβαια να αφήνουμε κατά μέρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βερσιά. Δύο ακόμη συναδελφοί που δεν είναι σκιώδης. Κυρία Κιλνίσλσεν πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταβάρες, σκιώδης ηγητής, αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αλλά θα ήθελα δύο λόγια μόνο πολύ σύντομα για να πω ότι είναι πολύ καλή έκθεση για μας, πληρέστατη, πλούσια σε υλικό, σε περιεχόμενο και Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, σκέψεις που διατυπώνονται προς τις ε, στρατηγικές εφαρμογές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ανθρώπινα δικαιώματα, ότι μας βρίσκουν σύμφωνους και θα την υποστηρίξουμε όπως είπα την έκθεση με μεγάλη χαρά. Κυρία Ντεκεζέ, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει πως φυσικά να πω ότι θα στηρίξω την έκθεση του συναδέλφου Χόβιτ, ούτε ότι δεν είναι εξαιρετή έκθεση. Πάντα παρακολουθώ κάθε χρόνο δηλαδή τις εκθέσεις αυτές και τις εξελίξεις στα ανθρώπινα δικαιώματα προς αυτήν την επιτροπή μας, τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα προς τους μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορούμε να επιχειρήσουμε μια βελτίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα στις ε, διάφορες χώρες και ιδιαίτερα σε διάφορα σημεία της εκθέσεως όπου γίνεται αναφορά δηλαδή σε διεθνείς συμβάσεις, ε, συμφωνίες, ε, δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα φερειπίν σε εμπορικές συμφωνίες, γίνεται λόγος για περισσότερη συνοχή από ορισμένους, περισσότερη ε, υλοποίηση, εφαρμογή από άλλους. Μέσα το σημαντικό είναι η συνοχή, η συνέπεια στα όσα λέμε και σε, σε αυτά τα οποία αναλαμβάνουμε στις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Και βέβαια ό,τι κάνουν και οι επιτροπέ του Κοινοβουλίου. Είναι ΙΝΤΑ, ΑΦΕΤ, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει πάντα να έχουμε συνέπεια, να δείχνουμε συνεπή στάση στη συμπεριφορά μα στι ε, τοποθετήσεις μας για να δώσουμε μια επιπλέον μόχλευση στα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό, το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το είχα διμέρω ε, κοινοποιήσει τον κύριο Χόουιτ, θα τον παρακαλέσω ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει βέβαια, αλλά θα ήθελα πολύ πιο ξεκάθαρα να αναφερθεί η προστασία των παιδιών μάγων όπως ονομάζονται στην Αφρική. Παιδιών που ανακηρύσσονται σε μάγους, κατηγορούνται για μαγεία και με δεδομένη και την ε, δυσπραγία που προξενεί είτε η οικονομική κρίση είτε η πόλεμη κατηγορούνται λοιπόν ε, για ε, μαγεία, για, για μαύρη μαγεία εξορκίζονται, τα, πετάνε, τα εξορκίζουν, τα πετάνε στους δρόμους ε, Μερικέ φορέ τα σκοτώνουν ακόμα. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει πολύ για τα παιδιά στρατιώτες, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και τα παιδιά μάγους που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα στην Αφρική. Ευχαριστώ και τελευταία ομιλήτρια ή αντιπρόεδρος παρακαλώ. Κύριε Σάντσιν Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ θερμά τον ε, Ρίτσαρτ για την πολύ καλή έκθεση. Δεν έχω καμία επιφύλαξη. Αναφέρεται το ζήτημα των ε, παιδιών αυτών. Ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μερικά σημεία. στο σημείο 81 Φερρυπίν, στη δουλειά που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα μπορούσαμε να ε, υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη για επαγρύπνηση. Θα αποτελούσε μια χρήσιμη όθηση για τη δουλειά που γίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα μπορούσαμε ως εκ τούτου να εξασφαλίσουμε έναν σαφέστερο και πιο ισχυρό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον αγώνα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριος Κλούπος, να από την Πολωνία, το είπε άλλωστε. Αναφερόμενο στο σημείο 64 ότι αυτό θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε και σε σχέση με τις ψυχικές ασθένειες. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να επιδιώξουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που γίνεται σε κράτη μη δημοκρατικά συνήθως. Θέλουμε ψυχικές ασθένειες να μην μπορούν να αξιοποιηθούν από ορισμένα καθεστώτα εις βάρος των ίδιων των ασθενών. Για να επιδεινωθεί δηλαδή η κατάσταση τους, η προστασία των δικαιωμάτων τους. Επίσης κάτι άλλο, πολύ συχνά κάνουμε λόγο για τη βία εις βάρος των γυναικών. Πολύ σωστά. Στην έκθεση έχει γίνει σχετική αναφορά, όμως θα ήθελα να επισημάνω και το εξή. Ότι ε, υπάρχουν κράτη που γνωρίζουν την απόλυτη απαγόρευση της άμβλωσης, ενώ κάποια άλλα τα οποία επιβάλλουν υποχρεωτική άμβλωση σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτά αποτελούν διάκριση εις βάρος των γυναικών και άρα θα πρέπει να αγωνιστούμε κατά και των δύο αυτών τύπων πρακτικών. Και τη απαγόρευση τη άμβλωση, γιατί και αυτή είναι διακριτική μεταχείριση βάρο των γυναικών, αλλά και τη υποχρεωτική άμβλωση. Γιατί πάλι η απόφαση για το άμβλωση ή μη ανήκει μόνο και μόνο στη γυναίκα την ίδια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Ακούσαμε, πιστεύω, όλου του συναδέλφου. Και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σβάνα από το ΕΑΕΣ, από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό που είπε και ο κύριος Χόουιτ το ίδιο, ότι δεν ήταν σε θέση να ε, μελετήσει τα έγγραφα από το διάλογο με την Κίνα και τη Ρωσία. Και όταν ήμουνα ένας απλός βουλευτής πέρσι, θυμάμαι, είχα πάει σε ένα δωμάτιο της υπηρεσίας εξωτερική δράσης ως απλός βουλευτής χωρίς βέβαια ούτε τσάντα ούτε μολύβι στα χέρια μου ε, σε ένα κλειστό δωμάτιο λοιπόν τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση μπόρεσα να διαβάσω τέτοια έγγραφα. Δεν ξέρω γιατί να άλλαξε αυτό εφέτο. Επίση λέτε ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι πιο περιορισμένη η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην δράση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Κύριε Σφόν, παρακαλώ. Thank you very much. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Προσπαθούσα να στείλω ένα μήνυμα για να μου επιβεβαιώσουν οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο αυτό σημείο της πληροφορίας, δηλαδή τη δυνατότητα πρόσβασης της πληροφορίας, γι' αυτό καθυστέρησα να λάβω το λόγο. Ε, διότι τουλάχιστον οριζοντίως δεν έχει γίνει αλλαγή πολιτικής, εξ όσων γνωρίζω. μάλλον. Είναι ξεκάθαρη η θέση του Κορεπέρ για την πρόσβαση στις πληροφορίες, βάσει της οποίας, μέσα στο πλαίσιο της οποίας εργαζόμαστε εδώ και το καιρό πια. Και δεν αφορά μόνο την υποεπιτροπή σας, αλλά και τη σχέση Συμβουλίου-Κοινοβουλίου εν γέννη. ως προς την ανάμειξη της ε, γραμματείας της Επιτροπής ε, στην προετοιμασία της εκθέσεως και πάλι δεν ξέρω ποια είναι η βάση για τα σχόλια αυτά, αφού είχαμε ετοιμάσει την ε, τορνή αλλά και την προηγούμενη έκθεση, αφού ετοιμάστηκε μάλλον η τορνή και η προηγούμενη έκθεση, από τις υπηρεσίες μας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ακολουθήθηκε η ίδια ακριβώς μέθοδος και ότι ε, ε, εξώσον εγώ γνωρίζω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πολύ ευχαρίστω όμως να εξετάσω περαιτέρω το πράγματα. Εν γέννη, θα έλεγα ότι η αιτήσια έκθεση ήταν πάντα συνεργατική μεταξύ Συμβουλίου Επιτροπής Κοινοβουλίου και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Ως βάση μου θα χρησιμοποιήσω την κοινή ανακοίνωση που ήταν και το αντικείμενο της προηγούμενης εκθέσεως. Και αν μου επιτρέπετε θα τη διαβάσω. Προκειμένου τη ασφαλιστή πρόοδο στην επίτευξη των στόχων προσδιορίζονται στην ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει την έκθεση πρόοδου τη μέσα στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ευρωπαϊκή πολιτική φορεί, συμπεριλαμβανομένε και τη κοινωνία των πολιτών, να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δράσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσδιορίσουν μελλοντικέ προτεραιότητε. Άρα το η τρέχουσα έκθεση συντάχθηκε, ετοιμάστηκε σε ένα έγγραφο περιγραφικό. Και αυτό γιατί το Συμβούλιο θέλησε μέχρι τώρα να έχει αυτό το αυτή τη διαμόρφωση του έγγραφου. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι από εδώ και μπρος βλέπουμε πως ε, τίθεται σε διαφορετική και νέα βάση αυτή η αιτήσια έκθεση. Μέχρι τώρα την ετοίμαζε το Συμβούλιο, με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία, με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και αυτό που ορίζει η κοινή ανακοίνωση είναι ότι η ετήσια έκθεση θα πρέπει να μετατραπεί σε έκθεση προς το Κοινοβούλιο μάλλον, απευθείας, που θα προσμετρά μέσα από ορόσημα τις επιδόσεις σε σχέση με τις φιλοδοξίες που έχουν προσδοριστεί στην κοινή ανακοίνωση. Και αυτό νομίζω ότι ε, σημαίνει προσέγγιση μάλλον της, ε, των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ τη υπηρεσία εξωτερική δράση, μελών τη Επιτροπή σα, εάν θέλετε κάτι ακόμη να αλλάξει κάποια, για να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα στον τύπο της παρουσίασης. Αλλά κατά τα άλλα υπάρχει πρόθεση συνεργασίας. Η έκθεση του κύριου Χάουιτ είναι μια έκθεση πλήρης. Εκτεταμένη. Δεν θα μου έφτανε ο χρόνος που έχουμε έρθει δεκάμιση, για να σας παρουσιάσω όλες τα σημεία. Για κάποια επιμέρου σημεία μόνο θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ευρύτατη βάση συνεννόησης μεταξύ της υπηρεσία μας, τις δράσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς την σοβαρότητα, τη σημασία της αντιμετώπισης των βασανιστήριων, την προτεραιότητα των δράσεων στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο, πιστεύω λοιπόν ότι τίνουν προ την ίδια κατεύθυνση. Τα σχόλια της Επιτροπής ε, των Επιτροπών Ανάπτυξης και Γυναικών ε, για την ενσωμάτωση φέρει πίν ε, ειδικών τμήματων της αιτήσιας έκθεσης σε, στους τομείς του εμπορίου και των ανθρωπών δικαιωμάτων τα λαμβάνουμε υπόψη, τα σημειώνουμε και πολύ ευχαρίστως ε, λαμβάνουμε γνώση των σχολείων αυτών και επίσης λεπτομερώς σας μια λεπτομέρειες θα ήθελα να πω ότι στη διατύπωση της εκθέσεως διατυπώνεται έτοιμα για ιδιαίτερη μέρημνα Υπογραμμίζω λοιπόν ότι η ετήσια έκθεση αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ε, στην έκθεση γίνεται λόγος για εκδημοκρατισμό, υποστήριξη του εκδημοκρατισμού. Όμως εμείς έχουμε πολιτική υποστήριξη της δημοκρατίας, όχι του εκδημοκρατισμού. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω όσο και αν σας φαίνεται ίσον θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθεί να επιβάλλει ούτε να εξαγάγει κάποιο σύστημα. Προσπαθεί μόνο να στηρίξει τη δημοκρατία όπου αναπτύσσεται αυτή από τις ρίζες προς τα άνω. Σας ευχαριστώ καταλαβαίνω δεν μπορώ βεβαίως να σας κατηγορήσω ε, εσάς για το ότι δεν έχουν πρόσβαση στην αξιολόγηση ε, οι βουλευτές. Θα το δούμε αυτό όταν ε, δούμε πώς μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα τα θεσμικά όργανα. Τέλος, ε, πεστάλη επιστολή για να έχω εγώ μία εξαίρεση, χωρίς να είμαι εισηγήτρια. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε ίσως να απευθύνουμε άλλη μία επιστολή για να πάμε στην Κομισιόν ε, και να περάσουμε σήμερα με και... Ό, όχι, όχι, όχι, όχι. Λάβετε το λόγο, αλλά να σας υπενθυμίσω πως πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα στις 11.30 να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης αλλά καταλαβαίνω πως οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, θέλουν να κάνουν κάποια σχόλια. David. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι ως τον πιο σύντομος. Εξ ονόματος όλου του δικτύου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη συνεργασία και στις διμερείς επαφές και στην ε, διαβούλευση υπήρξε μια ειλικρίνεια. Η ίδια η έκθεση είναι πάρα πολύ φιλόδοξη, έχει και πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει για να απαντήσει τα γεγονότα του 2010 και να μην αγνοήσει όλα όσα συνέβησαν το 2011 και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όσον αφορά τις θεσμικές εξελίξεις. Οπότε νομίζω πως είναι μια έκθεση που κοιτάει οπωσδήποτε το μέλλον και βεβαίως ε, αντικατοπτρίζει και τις συζητήσεις εντός του Συμβουλίου. Να αναφέρω κάποια πράγματα που ανέφερε ο κύριο Χάουιτ και κάποια άλλα τα οποία πρέπει να ενισχυθούν. Πρώτα απ' όλα για τις εκστρατείε ε, τις λεγόμενες, γιατί ο Χάουιτ είπε πως είναι επιφυλακτικές η ΜΚΟ ε, και θέτει πολλά ερωτήματα για το πώς αποφασίζονται αυτά τα πράγματα και το τι σημαίνει για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα θέλαμε να τα διαλέγει αυτά κανείς με ένα καπρίτσιο τα θέματα. Θέλουμε να υπάρχει μια εμπειρογνωμοσύνη ε, σε σχέση με αυτή την απόφαση. Κατόπιν για το διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρατε τον αποτυχημένο αυτό μηχανισμό. Δεν ξέρω αποτυχημένος, αλλά οπωσδήποτε γίνεται κατάχρηση σε πολλές ε, περιπτώσεις. Και παρά το ότι δεν έχουν οπωσδήποτε αποτελέσματα αυτοί οι διάλογοι, ε, εξακολουθούν να έχουν θέση σε μια ευρύτερη πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την πολιτική γειτονία αναφέρθηκε η βαθιά δημοκρατία και η σημασία που έχει και τα ζητήματα μη διάκρισης. Ε, αυτό φαντάζομαι πως θεωρεί πως συμπεριλαμβάνονται και όλα τα πολιτιστικά δικαιώματα τα οποία αγνοούνται αυτή τη στιγμή. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα. Δύο πράγματα που πρέπει να ενισχυθούν ίσως στην έκθεση. Ένα για την Ένωση και τις εμπορικές συμφωνίες δεδομένου του ότι ε, θα έρθουν πολλές εμπορικές συμφωνίες φέτος στο Κοινοβούλιο πρώτα απ' όλα με το Τουρκμενιστάν που ελπίζουμε να πάει στην Ολομέλεια τους επόμενους μήνες και υπάρχει μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια υποβάθμισης της ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη, οπότε το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σαφές για την αξία της ρήτρα αυτής. Εφαρμόζεται με κακό τρόπο κτλ. Ναι, εντάξει, να βρεθεί άλλος τρόπος εφαρμογής, αλλά η αξία ε, πρέπει νομίζω να αναφέρεται σε όλες τις συμφωνίες και τέλος για το τι μπορεί να κάνει το ίδιο το κοινοβούλιο ε, το κομμάτι για τον ρόλο του κοινοβουλίου νομίζω μπορεί να ενισχυθεί λίγο περισσότερο ειδικά όσον αφορά το τι κάνει το κοινοβούλιο εκτός αυτής της επιτροπής για τη συνέχεια που δίνεται στα ψηφίσματα κτλ. οι στάσεις μπορούν να γίνουν εκεί πέρα θα επιστήσω την προσοχή σας στην επιστολή την οποία απευθύναμε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου επί τη ευκαιρία της ε, εκλογής του. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω τον λόγο στον Ρίτσαρντ ε, με τις 99 παραγράφους. Α, κοιτάξτε, αν λάβετε υπόψη όλα όσα ακούστηκαν θα έχουμε 101 παραγράφους Ευχαριστώ. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της και η δική του παρουσίαση ήταν εκτενής. Αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί φιλοφρόνηση, το δέχομαι. Θα ήθελα να πω στους Σκιώδης, να ευχαριστήσω τους Σκιώδης για τη συνεργασία και πιστεύω ότι το κείμενο μπορεί να εγκριθεί. Θέλω να συνεργαστούμε για τροπολογίες και σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας εκ των προτέρων. Θα ήθελα να πω στην κυρία Σεντσίν και στη συνάδελφο εδώ δίπλα που ε, χαίρομαι, ότι χαίρομαι επειδή συνεισέφεραν, συνεισέφεραν και από την δική μου ομάδα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα θα απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με τα στοιχεία του κυρίου Τζιπ. Τα όσα ανέφερε, πιστεύω ότι ναι, θα πρέπει να δούμε όλα τα αντικειμενικά στοιχεία και τις πηγές και τα στοιχεία από πηγές. Δέχομαι αυτά που είπατε ως προς αυτά και εσείς ε, μιλήσατε για ε, εμπειρικά στοιχεία και για εμπειρογνώμα στοιχεία εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε όταν υπάρχει ασάφεια να τη διορθώνουμε. Εάν θέλετε ε, να μου πείτε για στοιχεία που δεν είναι ακριβή, να μου το πείτε μετά τη συνεδρίαση. Κατέβαλα κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσω να τεκμηριώσω τα στοιχεία που παρουσιάζω. Αν υπάρχουν κενά να μου τα πείτε στο τέλος. Ως προς τις ιδιαιτερότητες ε, και τον εκτενή χαρακτήρα comprehensiveness έκανα ό,τι μπορούσα για να φτάσω σε μία ισορροπία και αν ο κύριος Ζιπ θέλει κάτι να μου πει ε, όλες του οι παρατηρήσεις είναι πρόσδεκτες ως προς τη μεθοδολογία. Πιστεύω ότι υπάρχει μεθοδολογία και πρέπει να πούμε ότι στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνανε επικαλύψεις αναφερόμενοι χώρα προς χώρα. Νομίζω ότι λάβαμε μία απόφαση πέντε χρόνια πριν να μην το κάνουμε και ότι το Συμβούλιο θα, είναι, θα ε, αποτιμά την κατάσταση στην ετήσια έκθεση και εμείς θα κάνουμε μία αξιολόγηση. Εγώ ακολούθησα αυτή τη μεθολογία, γι' αυτό και το κείμενό μου... Το κείμενο μπορεί να είναι θεωρητικό, να φέρεται κάπως αφηρημένο και γι' αυτό δεν ορίζω πάντα τις χώρες προέλευσης. Ε, το λέω αυτό γιατί το είχαμε αποφασίσει στην Υποεπιτροπή. Θα ήθελα να πω στους κοιόδης, ως προς τροπολογίες, να μην μου στείλετε τροπολογίες αναχώρα. Δεν εργαζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο στην έκθεσή μας και ζητώ τη συνεργασία σας ως προς αυτό, έτσι ώστε να παραμείνουμε σε αυτή την αρχή, γιατί ε, αλλιώς υποτιμούμε τα δικά μας ε, δεδομένα. Ως προς τα τρία σημεία του κυρίου Τζιπ, για περισσότερο διάλογο με διεθνείς οργανώσεις ως προς τα, τη μετάβαση, τη μεταβατική περίοδο των χωρών της Αραβικής Άνοιξης, καθώς και το θέμα των θυμάτων. Ε, είναι ευπρόσδεκτες παρατηρήσεις του και θα περιμένω τις τροπολογίες σας. Ως προς τα θέματα που έφυξε η κυρία Βερζιά στο, ως προς το ίδιο θέμα, ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν παραποιήσεις, μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επικεντρωθούμε σε αυτά. Αν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη, είναι ευπρόσδεκτη. Όπως είπα στην κυρία Βερσιά και στην ΚΟΕ, μας ενδιαφέρει να ε, έχουμε μία αξιολόγηση ε, και δέχουμε το mainstreaming που προβάλλεται. Προς την κυρία Ντεκεζέρ θα ήθελα να πω ότι τα σημεία που αναφέρει με βρίσκουν σύμφωνο ως προς τις διεθνείς συμφωνίες, τις δηλώσεις αντικτύπου, και σε ένα προωθημένο στάδιο αποφάσεων. Θα ήθελα να δείτε αυτά τα ορόσημα και να μου πείτε αν εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και να κάνουμε συστάσεις. Θα ήθελα να ε, μου δώσετε στοιχεία υπομορφή ανάδρασης ως προς την αντιμετώπιση των ανηλίκων θα πρέπει σε αυτή την παράγραφο να εντάξουμε και άλλα στοιχεία. Στην κυρία Σέντσιν θα ήθελα να πω ότι σε προηγούμενες εκθέσεις μιλήσαμε ε, για τα πρόσωπα, για τα άτομα με, με ειδικές ανάγκες, προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα μαθησιακά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε ένα τόσο λεπτό θέμα υπ' αυτή τη μορφή, επειδή ασχοληθήκαμε με θέματα ε, ειδικών αναγκών, σε άλλες εκθέσεις θα πρέπει να δούμε κατά πόσο εδώ το θέμα είναι πιο επικεντρωμένο. Μπορείτε να προετοιμάσετε ε, μία τροπολογία. Ο κύριος Τσίπ μίλησε για σεξουαλικό προσανατολισμό στην παράγραφο 64. Γνωρίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα, ιδιαίτερα για το ΕΛΚ, αλλά είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας για μένα και την ομάδα μου, καθώς και για πολλούς άλλους. ως προς την κακή ιατρική διάγνωση για να αρνηθούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων ως προς το σεξουαλικό τους προσανατολισμό πιστεύω ότι το θέμα αυτό μπορεί να τύχει συμφωνίες. Δεν θα πρέπει να έχουμε εσωτερικούς διχασμούς, γι' αυτό και έθιξα αυτό το θέμα. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Κατανοώ ε, ότι υπάρχει μία ευαισθητοποίηση από την ομάδα του κυρίου Τζιπ, γι' αυτό να δούμε πώς μπορούμε Ας δούμε πώς μπορούμε να το διαρθρώσουμε, να το εκφράσουμε γλωσσικά για να φτάσουμε σε συμφωνία. Σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία νομίζω ότι μπορούμε να διορθώσουμε το κείμενο, το βελτιώσουμε. Με ενδιαφέρει έλλειψη διακρίσεων και δέχομαι αυτά που είπατε ως προς τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ίσως σε θέματα ορισμένων χωρών, Ινδίας και Καναδά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να εντάσσεται σε κάθε συμφωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένες χώρες σε αυτόν τον κατάλογο, εάν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν έχω διαβάσει αυτή την επιστολή προς τον πρόεδρο Σούλτς. Αν ε, θεωρείται εμπιστευτικού χαρακτήρα το, το έγγραφο αυτό, την επιστολή, ε, τότε θα σας υποσχεθώ ότι δεν θα ε, διαβιβάσω αυτά τα στοιχεία σε κανέναν προς τον ε, κύριο Σβάν θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Ε, το είχαμε κάτι ε, επί του θέματος και νομίζω ε, ότι κάνουμε μία μικρή πρόοδο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι είναι μία μακροχρόνια διαδικασία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και πρόοδος. Όταν μιλώ για failed mechanisms, δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύω στο διάλογο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές φορές όμως υπολοιπόμαστε σε σχέση με τις προσδοκίες μας και ίσως θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ε, θα προχωρήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Κύριε Σουάν, πέρα από τις διαφωνίες του παρελθόντος θα πρέπει να έχουμε μία αξιολόγηση με βάση την αποτελεσματικότητα. Δέχομαι ε, αυτή την ε, προσέγγιση σε σχέση με το παρελθόν. Ως προς δημοκρατία και τον εκδημοκρατισμό, νομίζω ότι, οι ε, κύριε Σουάν, υπήρχαν συμπεράσματα του Συμβουλίου επί του θέματος. Θα πρέπει να ανατρέξουμε στο παρελθόν, κύριε Σουάν. Για λόγους ε, χρονικής, οικονομίας χρόνου δεν μπορέσατε να επεκταθείτε, αλλά θα ήθελα τα γραπτά σας ε, σχόλια σε σχέση με ε, επιμέρους ζητήματα που άπτονται της δραστηριότητας της ΕΕΔ. Μπορείτε να μου κάνετε λοιπόν και γραπτές υποδείξεις έτσι ώστε να διασαφίσω ορισμένα σημεία του κειμένου εάν αυτό το κρίνουμε σκόπιμα. Ευχαριστούμε κυρία Χάουιτ. Ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Πρόθεσμοι για τροπολογίες είναι 15 Φεβρουαρίου, 6 ώρα το απόγευμα. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης. Ακρόαση για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Έχουμε εδώ πέρα εμπειρογνώμονες. Αυτή η ακρόαση γίνεται μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών. Αναμένουμε τον Πρόεδρο ακόμα, αλλά ορίζω τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και αυτό γίνεται από κοινού με την αντιπροσωπεία των χωρών μας ΡΕΚ και καλωσορίζουμε τον κύριο Ντέιβιτ. Τώρα η υποεπιτροπή μας ενημερώνεται τακτικά ακούγοντας ειδικού ε, της κοινωνίας των πολιτών από τις διάφορες χώρες για το πώς πάντα πράγματα. Οπότε είχαμε καλεσμένους από την Ιεμένη, τη Συρία και τώρα θα δούμε το τι γίνεται στην Αίγυπτο. Και πριν ξεκινήσουμε, νομίζω πως όλοι γνωρίζουμε τις φρικτές εικόνες που είδαμε μετά το, τον ποδοσφαιρικό αγώνα στο Port Said και βεβαίω συλληπούμεθα τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά οπωσδήποτε το πολιτικό αίτημα είναι μια ανεξάρτητη έρευνα για το ποιο είναι υπεύθυνο. Βεβαίω, πάντα δημιουργούν προβλήματα οι οπαδοί, αλλά εάν δεν αντιδράει η αστυνομία... Uh, fight between two soccer games, soccer groups. Ε, μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα μεταξύ διαφόρων ομάδων, οπαδών. Επίσης υπάρχει καταστολή των ΜΚΟ και των διεθνών ΜΚΟ και ο Πέτερινγκ αυτή τη στιγμή είναι στην Αίγυπτο για να παρακολουθήσει κάποιες τέτοιες ε, περιπτώσεις γιατί είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Adenauer από το οποίο επίσης έχουμε εκπροσώπους οπότε νομίζω πως Τώρα θα ξεκινήσουμε, θα περιμένουμε τον κύριο Μπρόκ, όταν έρθει θα τον ακούσουμε, αλλά μετά θα γίνει και μια ακρόαση και κλεισμένο το θυρών για τη Ρωσία. Οπότε παρουσιάζω τώρα τους καλεσμένους μας. Είναι ο Αχμέτ Σαμί, διευθυντής του Ινστιτούτου Ανταλούς ε, στο Κάιρο, ο κύριος Ντβόρκιν, ο οποίος είναι συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων και καλώς ήρθατε και ο δόκτωρ Στέφαν Γκέρελ, διευθυντή του ε, Ευρωπαϊκού Γραφείου του Ιδρύματος Αντενάουερ και επίσης είχαμε και συστάσεις από τους ε, συναδέλφους για να έρθει κάποιος από την Human Rights Watch. Προσπαθήσαμε, αλλά η εκπρόσωπός τους ε, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή και δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί μαζί μας. Και από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι εδώ πέρα η κυρία Νασίρα Μπούλου, ε, η οποία είναι επικεφαλής της μονάδας για τη Μέση Ανατολή. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Σαμίρ, ο οποίος θα μπορούσε ίσως να περιοριστεί σε με 7 με 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι εκλογές μόλις ολοκληρώθηκαν για την Εθνοσυνέλευση, αλλά οι εκλογές ε, δεν σημαίνουν δημοκρατία, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς τα δικαιώματα των γυναικών. Καθώς βλέπουμε πως από 508 από 508 βουλευτές ε, οι γυναίκες δεν είναι καν 10 και πολλές από αυτές ε, διορίστηκαν όλες. Και πρέπει να υπάρχουν βεβαίως και ελεύθερα μήμυε. Σε μια χώρα δε όπου 40% του λαού είναι πολύ φτωχή, η δημοκρατία δεν ε, σημαίνει πως υπάρχει όταν ε, ένα-δύο πολιτικά κόμματα έχουν τεράστια οικονομικά μέσα. Κυρίες και κύριοι, ο Ζαν Ζακρουσό και το κοινωνικό, στο κοινωνικό, στο κοινωνικό συμβόλαιο μιλούσε βεβαίως για τη σχέση μεταξύ πολιτών και κρατών. Είναι σχέση ε, πατέρα και γιου. Στην Αίγυπτο βλέπω πως ο πατέρας δεν μπορεί να δεχτεί πως ο 25χρονος γιος του κάνει ό,τι θέλει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά και πολύ πολύπλοκα ταυτόχρονα. 75% του λαού της 65% ε, είναι κάτω από 25 ετών. 40% είναι και κάτω από 25 ετών. Και γνωρίζω πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θέτει αυτά τα ερωτήματα, το τι πρέπει να κάνουμε. Ο Τόμας Φρίντμαν είχε γράψει σε ένα μοναδικό άρθρο μετά μία επίσκεψή του στην Αίγυπτο πως όταν βλέπεις ελέφαντες να πετάνε σκάσε και κράτα σημειώσεις. Υπάρχει και ένας ε, Αιγύπτιος ε, διανοητής που είχε γράψει πριν από δύο μέρες, ναι, η Επανάσταση πέθανε, η Επανάσταση επέτυχε, η χώρα πέθανε. Εννοούσε ότι το παλαιό καθεστώς δεν μπορεί να ανανεώσει και να ξαναχτίσει αυτόν. Πολλοί νέοι Αιγύπτιοι Ε, μιλούσαν για μεταβατική περίοδο. Εμείς το λέγαμε περίοδο εκδίκησης. Καμία χώρα δεν ε, περνάει στην δημοκρατία όταν ε, συνασπίζονται οι στρατιωτικοί με τη μουσουλμανική αδελφότητα για να μην αλλάξει τίποτα. Και μετά την πρώτη εβδομάδα της Αιγυπτιακής Εθνοσυνέλευσης αντιλαμβάνεστε πως ε, λαμβάνει η χώρα μία μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, το κόμμα Μουμπάρακ, ε, ε, έχει μετακινηθεί προς τους προς σαλαφιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Ναι, δεν είναι του πρώην καθεστώτος, αλλά δρούν ακριβώς όπως το παλαιό καθεστώς. Όταν βλέπετε τον Υπουργό Εσωτερικών, να αρνείται στην ε, Εθνοσυνέλευση το ότι χρησιμοποιήθηκαν πυροβολισμοί για να σταματήσουν τους διαδηλωτές. Και όταν βλέπετε βουλευτές να χειροκροτούν τις δηλώσεις αυτές, καταλαβαίνετε πως η διαφορά αφορά μόνο τα ονόματα και όχι την ουσία. Ειδικά όταν πολλές εκθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνείς και ε, τοπικές λένε πως η αστυνομία χρησιμοποιεί τη μέγιστη βία για να σταματήσει τους διαδηλωτές. Δεν ε, μπορούμε να ζητήσουμε από έναν ε, γραφειοκράτη ή στρατηγό να χαράξει το μέλλον της Αιγύπτου και εάν η κατάσταση παραμείνει τόσο σκοτεινή προτείνω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην στήριξει αυτό το καθεστώς. Το Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει πρόβλημα νομιμοποίησης και η κυβέρνηση επίσης. Και όταν τα περισσότερα πολιτικά κόμματα κάθε μέρα εκθέτουν ε, αυτούς και το κοινοβούλιο χάνουν την νομοποίησή τους και όταν δείτε την οργή της ε, πραγματικής πλειοψηφίας, δηλαδή των νέων στους δρόμους, η κατάσταση είναι ασταθής. Ακόμα και αν ήθελε κανείς να στηρίξει μια κυβέρνηση, βλέπουμε πως ε, μιλάμε για στενόμυαλες πολιτικές ομάδες, ειδικά οι σαλαφιστές και η μουσουλμανική αδελφότητα, η αδελφή μουσουλμάνια. Όταν η ΜΚΟ της Αιγύπτου και οι διεθνείς αντιμετωπίζουν συνεχείς επιθέσεις από την κυβέρνηση και το στρατό και το κοινοβούλιο γιατί κατά βάση κάνουν τη δουλειά τους όταν τους κατηγορούν συνέχεια ότι είναι πράκτορες της Δύσης here in τότε τι δημοκρατία έχουμε στην ε, Αίγυπτο, τι μέλλον μπορούμε να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο συνέβη στο Port Said δεν ήταν χουλιγανισμός. Οι διαφορετικές ε, διερευνητικές αποστολές έδειξαν πως υπήρχε στόχευση συγκεκριμένου ακτιβιστή που ήταν σε μια ομάδα οπαδών που ήταν κατά του στρατού και του ανωτάτου στρατιωτικού συμβουλίου. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube που το δείχνουν. Και κυρίε και κύριοι, όταν ο Αιγυπτιακός στρατός χρησιμοποιεί τη μέγιστη δυνατή βία σε σημείο να σκοτώνει διαδηλωτέ και να να ξεγυμνώνει γυναίκες διαδηλωτές στους δρόμους του Καΐρου τι περιμένετε να κάνει ε, τι εγγύηση μπορεί να έχει η νέα γενιά της χώρας μου από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει μια ιστοσελίδα που λέγεται scafcrime.net και .com ε, που δημιουργούν οι διάφοροι blogger της Αιγύπτου πήγαινε εκεί πέρα να δείτε με στοιχεία εικόνες και βίντεο το τι γίνεται στους δρόμους ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Σάμι, για τα λόγια σας. Και μάλιστα μου θυμήσατε μια συζήτηση που έγινε χθε στην ΑΦΕΤ για τη Ρωσία. Ακριβώς το ίδια επιχειρήματα. Οι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις παίρνουν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποιοι δηλαδή οι οποίοι προσπαθούν να ε, αποσταθρώσουν την νομοποίηση του έργου των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και επίση θα ήθελα να πω, γιατί λησμόνισα θα το πω στην αρχή, ότι η κατάσταση είναι πολύ κακή, επιδεινώνεται, αλλά ταυτόχρονα με ικανοποίηση χαιρετίζουμε την απελευθέρωση, αποφυλάκηση του blogger Mike Nabil. Είναι ένα καλό δείγμα. Νομίζω ότι και η διεθνή αλληλεγγύη συνέβαλε στην αποφυλάξη αυτή. Ο κύριος Δουόρκινγκ τώρα παρακαλώ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Επιτρέψτε μου σας τη δική μου προοπτική για την ε, κατάσταση στην Αίγυπτο και τη σημασία βέβαια των εκλογών και της μετακλογικής περίοδου. Η διεξαγωγή γενικών εκλογών και εκλογών νομίζω ήταν σημαντικό ορόσημο στις εξελίξεις που θα χαρακτηρίζω ως μεταλλαγή στην ε, Αίγυπτο, ίσως το σημαντικότερο βήμα μετά την αποχώρηση του Πρόεδρου Μουμπάρακ. Εισάγει για πρώτη φορά μια ομάδα αντιπροσωπευτική μέσα στο Κοινοβούλιο που μπορεί να αντισταθεί, να βρεθεί αντιμέτωπη στην ΣΚΑΦ, δηλαδή στην, ε, στο Ελλοντατό Συμβούλιο των Ενωπλών Δυνάμεων πλην όμως, και όπως είπε και ο σα είναι ανεπαρκής, ατελής ε, αυτή η προσπάθεια. Να τελέσει το βήμα προς την μετάβαση στη δημοκρατία. Και έτσι αφήνει πίσω του μια κατάσταση συγκεχημένη, μια κατάσταση που δεν υπάρχει γενική συνένεση για τις περαιτέρω εξελίξεις του, του πολιτικού συστήματος, μια κατάσταση όπου δεν είναι σαφές πώς μπορεί να προκύψει συμφωνία μεταξύ μέσα στην πολιτική κοινωνία μεταξύ του πολιτικού προσωπικού της Αιγύπτου για να φτάσει σε μια πολιτική συνένεση η χώρα που αποτελεί πιστεύω για μένα και το ουσιαδέστερο πρόκριμα μιας δημοκρατίας. Άρα λοιπόν έχουμε την αντιπαράθεση μεταξύ τη δηλαδή στρατιωτικής ηγεσία του Κοινοβουλίου στο οποίο επικρατούν οι αδελφοί μουσουλμάνοι και των διαδηλωτών του κοινού, του απλού κόσμου στο δρόμο. Τρεις ομάδες λοιπόν, από των οποίων καμία δεν έχει ξεκάθαρη νομοποίηση αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει αυτή η διεκδίκηση της νομοποίησης που διαπιστώνουμε τώρα. Το κόμμα της ε, ελευθερίας και της δικαιοσύνης των αδελφών μουσουλμάνων στο Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ο ρόλος του είναι μια κατεκχώρηση εξουσία, έχει εκλεγεί πλέον και θεωρεί ότι είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με την στρατιωτική ηγεσία χωρίς να λαμβάνει πλέον υπόψη του την συμμετοχή του λαού στην πολιτική, στο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν υποστηρίζει πλέον τους διαδηλωτές, θέλουν να σταματήσουν αυτές τις διαδηλώσεις, δηλαδή και κλεισμένων των θυρών να αναπτύξει μια σχέση με τη στρατιωτική ηγεσία. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ε, προσπάθειες ε, για ε, διαπραγμάτευση μιας γενικής αμνηστίας με την στρατιωτική ηγεσία που όμως απέτυχε παταγωδός και δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Ο κύριος Σάμι νομίζω μίλησε εύκολα για τις παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων που σημειώνονται στην Αίγυπτο. Ένα ζήτημα που θα ήθελα και εγώ να προσθέσω θα ήταν η διάσταση του μέλλοντος, να κοιτάξουμε μπροστά. Και τώρα μπροστά μας έχουμε τη συνταγματική διαδικασία. Ε, το χρονοδιάγραμμα, ο δικός χάρτης ε, που έχουμε δείχνει ε, διατύπωση και έγκριση νέου συντάγματος πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες προεδρικές εκλογές προβλέπονται για τις αρχές Ιουλίου ή και νωρίτερα. Άρα δεν αφήνει περιθώριο το χρονοδιάγραμμα αυτό για μια διαδικασία ομαλή τακτική που θα επέτρεπε την ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου όπως αυτός απαιτείται για την ανάπτυξη της πολιτικής συνένεσης και διευθέτησης. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται είναι μάλλον μια ε, κατεπίγουσα διαδικασία εισαγωγή νέου συντάγματος ή επιδιόρθωσης του παλαιού συντάγματος του 1971 και έγκρισής του και έτσι πιστεύω ότι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο ανησυχία στο δρόμο για μια νέα πολιτική διευθέτηση που περιμένουμε με αδημόνια στην Αίγυπτο. Επίσης, οι εξουσίες του Κοινοβουλίου, του Ανακλήκεντος Κοινοβουλίου, έχει νομοθετικές εξουσίες με βάση τον διάμεσο, το μισοπρόθεσμο συντάγμα, που θέσπισαν οι στρατιωτικές αρχές, δεν διαθέτει τέτοιου είδους εξουσίες και όμως στο Κοινοβούλιο διεκδικεί νομοθετικές ουσίες. Ταυτόχρονα όμως και παράλληλα, όπως επεσήμανε και ο κύριος Σάμι, το ΣΚΑΦ, η στρατιωτική ηγεσία, ξεκολουθεί να κυβερνάει τη χώρα χωρίς ανοχή καμία, ε, χωρίς πλουραλισμό κανένα και χωρίς ε, ένδειξη ότι σκοπεύει να στραφεί προς τη δημοκρατία. Έχουμε περιστολή των δικαιωμάτων των μαζικής ενημέρωσης, ε, καθεστώς έκτη της ανάγκης, στρατοδικία, καταστολής της μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και έτσι η στρατιωτική ηγεσία φαίνεται ότι ε, συλλέγοντας πληροφορίες από την υπηρεσία πληροφοριών ε, ε, προσπαθεί να δίνει την εντύπωση ότι υπάρχουν ε, συνωμοσίες έξωθεν για την καταστολή των ε, των ε, διαδηλώσεων και εδώ έρχεται το ζήτημα της χρηματοδότησης από πλευράς των ΗΠΑ των διαδηλωτών ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων που οργανώνουν τις διαδηλώσεις. Υπάρχουν ζητήματα βέβαια ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είδαμε ότι δεν ήταν δυνατή η διατήρηση της τάξης και ασφάλειας σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Άρα είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες ε, για τον έξω κόσμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει βέβαια να υποστηρίξει την ε, μετάβαση στη δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνει και κίνδυνο η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρηθεί παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να επικεντρωθούμε στο σωστό μήνυμα, δημόσιο μήνυμα που θα αποσταλεί για να εξασφαλιστεί μέχρι τη δυνατή νόμιμοποίηση στα νέα δεδομένα στην Αίγυπτο και τον προσδορισμό των νέων και κύριων προτεραιοτήτων. Ένα είναι το μήνυμα, πιστεύω. Ένα πρέπει να είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη στηρίζει τις ε, προσδοκίες του Αιγυπτιακού λαού, δεν προσπαθεί να επιβάλλει δικό της πρόγραμμα η ατζέντα, στηρίζει τις προσδοκίες και διεκδικήσεις του Αιγυπτιακού ε, λαού για μια διαδικασία πολιτική, δημοκρατική, ισότιμη, πλουραλιστική, με σεβασμό του κράτους δικαίου και των βασικών ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου και πιστεύω ότι η πολιτική διαδικασία, η σταγματική διαδικασία πρέπει να είναι ε, ε ανοιχτή σε όλους, να στηρίζει το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις αρχές και ελευθερίες που γράφονται στο επίκεντρο της Νέας Δημοκρατικής Διαδικασίας. Στην οποία βέβαια έχει ρόλο η κοινωνία των πολιτών. Είναι λεπτή ισορροπία όντως. Ωστόσο η δήλωση του, της είπα της εκπροσώπου ως προς την ε, καταστολή αυτή στο ποδοσφαιρικό αγώνα ήταν μάλλον ατυχής γιατί έκανε λόγο για τήρηση των διαδικασιών. Πλην όμως εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε να κάνουμε με κατάχρηση υφισταμένων και άδικων νόμων, κατα... Ε, κατασταλτικών νόμων και άρα θα έπρεπε αντί για τήρηση των ε, νομικών διαδικασιών ε, να γίνεται λόγος μάλλον για Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν, για πλουραλισμό. Ε, κύριες προτεραιότητες ε, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα πλαίσιο για μια νομιμοποιημένη κυβέρνηση, πλουραστική κυβέρνηση, στηριζόμενη σε πολιτική συνένεση, διαπραγμάτευση και συνένεση με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βόρκιν για, την, για τις δηλώσεις σας και τις συστάσεις σας. Ο Δόκτωρ Γκέραλτ έχει τώρα το λόγο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Ιδρύματος Adenauer. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για το ότι με προσκαλέσατε. Είπαμε πως έχω 7 με 10 λεπτά να μιλήσω Να σας πω πως ως ε, διευθυντής του γραφείου Conrad Adenauer δεν είμαι ειδικό για τον αραβικό χώρο. Είχα δραστηριοποιηθεί στη Δυτική Αφρική και Θα ήθελα να παρουσιάσω λοιπόν την ε, άποψή μας ε, τη σημερινή. Θα αναφερθώ σε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα την το τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής ε, στο γραφείο μας ε, στο Κάιρο, δεύτερον ε, ποιους εταίρους έχουμε εκεί πέρα και τρίτον τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Κυρίε και κύριοι, το Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο εδώ και 30 χρόνια και συνεργάζεται με διάφορες οργανώσεις μη κυβερνητικές και με την κυβέρνηση και με τις επιχειρήσεις. Έχουμε έναν παγκόσμιο στόχο που είναι η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη των δημοκρατικών δομών. Ο συναλφός μου εκεί πέρα, ο δόκτωρας Ιάκοψ, είναι ειδικό στο Ισλάμ. Ε, σπούδασε πολιτικές επιστήμες ε, και Ισλαμικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της ε, Κολονίας ε, και πρέπει να πούμε επίσης πως είναι παντρεμένος και έχει εκεί πέρα δύο μικρά παιδιά οπότε η κατάσταση νομίζω τον αφορά και προσωπικά. Τώρα, λίγα λόγια για τις εξελίξεις. 29 12 του πέρσι το γραφείο του Ιδρύματός μας ερευνήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, την αστυνομία, ε, κατόπιν εισαγγελική ε, παραγγελίας, χωρίς όμως να μας επιδείξουν ένταλμα. Διάφορα έγγραφα και όλοι μας οι υπολογιστές ε, κατασχέθηκαν και σφραγίστηκαν τα δωμάτια και μας απαγορεύθηκε μέχρι νεοτέρας να συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας. Ε, τρεις πρώτου του 2012 κατόπιν προσεκλήθη ο κύριος Γιάκομπς και ανακρίθηκε για 5,5 ώρες από τον ανακριτή για να απαντήσει για τις κατηγορίες που βάριναν τον ίδιο και το Ίδρυμα. Του υποσχέθηκαν πως θα μπορέσει να επαναλάβει τη λειτουργία του το Ίδρυμα και θα του επιστραφούν τα έγγραφα και ο εξοπλισμός. Στις 11 Ιανουαρίου η εισαγγελία μας ενημέρωσε πως θα συνεχιστεί η δίκη και πως τα έγγραφα και οι υπολογιστές ε, κατάσχονται, μάλλον παραμένουν κατασχεμένα. Ο καθηγητής ε, ο κύριος Πέτερινγκ, ε, πρόεδρος του Ιδρύματός μας και πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, θεώρησε αφαίρετες αυτές τις ενέργειες. 18 πρώτου, ο Γενικός Γραμματέας του Τσεντεού, ο κύριος Γκρουλ, ίσως τον ξέρετε, ξέρετε πως δεν εξαρτώμεθα οικονομικά από τους Γερμανούς χριστιανοδημοκράτες αλλά συνδεόμαστε ιδεολογικά. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Αιγύπτιο πρέσβη στο Βερολίνο και είπε πως η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών εξαρτάται και από την ελεύθερη δράση μη κυβερνητικών οργανώσεων και ειδικά του Ιδρύματος Κόνραντ Άντενάουερ. 31ου Πήγε ο Υπουργό Εξωτερικών ο κύριος Βέλε, στο Κάιρο και συναντήθηκε εκεί πέρα με τις αρχές και έθεσε το ζήτημα της εργασίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων, άσκησε κριτική ε, στην ε, συμπεριφορά των Αιγυπτιακών ε, Αρχών και 5 Δευτέρου αυτή την εβδομάδα η εισαγγελία μας ενημέρωσε πως τώρα θα ξεκινήσει ποινική διαδικασία κατά του δόκτωρος Γιάκομπς και της κυρίας Μπάντε υπαλλήλου και στους δύο έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα ταυτόχρονα καταδίκασε σε συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρέσβη, τον κύριο Ράμζη, ο κύριος Πέτερινγκ αυτές τις δράσεις. Χτες το βράδυ ο δόκτωρ Πέτερινγκ πήγε στο Κάιρο και συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών και την Υπουργό Διεθνών Σχέσεων. Περνάω τώρα στο δεύτερο μέρος, το θέμα των κατηγοριών. Υπάρχουν δύο ε, τομείς ε, δραστηριοτήτων που μας αφορούν. Το ένα αφορά ζητήματα δημόσιας τάξης, δηλαδή το ένα είναι πως λειτουργούμε παράνομα ως ΜΚΟ στη χώρα και η δεύτερη κατηγορία είναι πως εξ, εξίσου παράνομα χρηματοδοτούμαστε με χρήματα από το εξωτερικό χωρίς να υπάρχει καταγραφή στη χώρα και εργάζονται επίσης αδήλωτοι εργαζόμενοι στη χώρα. Ε, πρόκειται για κατηγορίες εναντίον του Ιδρύματος και του Δόκτρος Γιάκοψο εκπροσώπου του Ιδρύματος και τώρα έχουμε και την ε, επιπλέον κατηγορία, έχουμε μάλλον την ποινική διαδικασία η οποία ξεκίνησε, δεν ξέρουμε ακριβώς ε, γιατί όμως θα κατηγορηθεί τελικά ο κύριος Γιάκομψο, μπορεί να είναι πράγματα όπως η κατασκοπία ή η προδοσία αλλά δεν, δεν το ξέρουμε γιατί δεν μας έχουν δώσει ακόμα τα έγγραφά μας. Το έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνει αυτό τις επόμενες τρεις ημέρες. η ε, δε ε, συνεταίροι του Ιδρύματος να σας πω πως κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ανακοινώθηκε στον δόκτωρα Γιάκομπς πως δεν ασκείται κριτική στη συνεργασία του με Αιγυπτιακές ΜΚΟ, αλλά υπάρχει εδώ πέρα ένας μικρός κατάλογος ε, εταίρων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Είναι το Κέντρο Στήριξης ε, Αποφάσεων, ένα ερευνητικό ίδρυμα ε, του Υπουργικού Συμβουλίου της Αιγύπτου, κατόπιν το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, το Κέντρο Οικονομικής Έρευνας και Μελετών, το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και Μελετών, Συνεταίρη στην ανάπτυξη, αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις γυναίκες και τα παιδιά, Al Sadat για την κοινωνική ανάπτυξη και Αιγυπτιακό Ίδρυμα νεολαία. Αυτή είναι η εταίροι του ε, Ιδρύματος στην χώρα. Έρχομαι τώρα στο τρίτο θέμα. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σήμερα στην Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή συζητείται αίτημα του Τσέντεου Τσέσου και του FDP για να απασχολήσει το θέμα αυτό τη Βουλή. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω ολόκληρο το αίτημα, μόνο τα σημαντικότερα σημεία. Ε, λέει το εξής. Ζητάει το Κοινοβούλιο από την γερμανική κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα η δίωξη εις βάρος του Ιδρύματος Κόνραντ ε, να επιτραπεί η λειτουργία των ΜΚΟ και να αναγνωριστεί η σημασία τους για την διαδικασία δημοκρατικού μετασχηματισμού και τρίτον πρέπει να ξεκαθαρίσει το ότι για την ε, Γερμανία έχει μεγάλη σημασία η ελεύθερη δραστηριοποίηση των γερμανικών πολιτικών ίδρυμάτων και θα ήθελα να πω πως διμερός η Γερμανία διέγραψε 240 εκατομμύρια χρέους, ήθελε να το κάνει αυτό ως αποτέλεσμα της Αραβικής Άνοιξης και επιπλέον διέτησε 140 εκατομμύρια για την ανάπτυξη της περιοχής, τα οποία θα ωφελήσουν και την Αίγυπτο. Να προσθέσω επίσης ακόμα πως ε, λογικό θα ήταν οι Αιγυπτιακές αρχές να λάβουν υπόψη πως το Δέλτα Σίγμα του Ιδρύματός μας είναι ο Χέλμουτ Κόλ, η κυρία Μέρκελ και ο πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο μέρος. Μπορώ να πω πως ε, δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή προς το καλύτερο της κατάστασης, μάλλον μία επιδίνωση. Ο κύριος Πέτερινγκ, ε, όπως είπα, θα συναντηθεί με τους υπουργούς. Οι αρχές ε, της Αιγύπτου υπενθυμίζουν και λένε πως δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση του Ιδρύματος Adenauer, αλλά πως πρόκειται για μία δίκη στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού συστήματος υπάρχει διάκριση των εξουσιών, δηλαδή η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δεν επηρεάζεται. Ένα τελευταίο ερώτημα. Αν πως πρέπει να φύγουμε από τη χώρα. Α, μάλλον όχι. Είμαστε δρεωμένοι στην Αίγυπτο και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εκεί και να πω πως για εμάς είναι άρα κάπως δύσκολο να ε, συνεχίσουμε την εργασία μας γιατί η κυρία Μπάντε η οποία επίσης κατηγορείται εκεί πέρα ε, είναι και αυτή παντρεμένη με Αιγύπτιο οπότε δεν μπορεί και αυτή να εγκαταλείψει έτσι απλά τη χώρα βεβαίω απειλείται με ποινική δίκτυο. σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας ευχαριστούμε κύριε Γκέρολτ για την παρουσίαση της κατάστασης ε, του τι συμβαίνει με το Ίδρυμα Adenauer είναι σοβαρή κατάσταση και βεβαίως εάν ένα τέτοιο Ίδρυμα που το αναφέρατε έχει τους δεσμούς με την Καγκελάριο και τους διαφόρους υπουργούς αντιμετωπίζεται έτσι ε, φανταστείτε τι κάνουν οι Αιγυπτιακές αρχές με μια τοπική μικιό που δεν έχει τέτοιους δεσμούς. Θα ήθελα τώρα πριν δώσω το λόγο στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ε, έχω μπερδευτεί με τους διάφορους δόκτορες εδώ πέρα. Λοιπόν, Γυρνώντας, ε, μιλώντας στα αγγλικά, θα ήθελα να ζητήσω από τον ε, κύριο Ντέιβιτ, ο οποίος ασχολείται με τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ, να μας πει και εκείνος, να μας δώσει και εκείνος μερικά στοιχεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και είμαι και ευγνώμων στα μέλη, προς τα μέλη του πάνελ που μας δώσανε μια σαφή εικόνα της πραγματικότητας για το τι συμβαίνει σήμερα στην Αίγυπτο. Το ζήτημα είναι κατά πόσο μας εκπλήσουν αυτά τα αποτελέσματα και νομίζω ότι η απάντηση είναι αρνητική από τους περισσότερους. Τα, εκλογικά αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα. Και επειδή είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορώ να ε, μιλήσω ελεύθερα, μπορώ να πω ότι όλα ήταν αναμενόμενα. Όσον αφορά την μουσουλμανική αδελφότητα, ε, είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ήμουν στην Αίγυπτο όταν ε, συζητήθηκε πρωταρχικά ο εκλογικός νόμος και μιλώντας με τις διάφορες πολιτικές ομάδες και εκπροσώπους διαφόρων ε, ιδεολογιών και επειδή ζούμε σε δημοκρατικές χώρες ευτυχώς και ζούμε σε δημοκρατικά εκλογικά συστήματα, μπορέσαμε να προβλέψουμε τα αποτελέσματα ενός τέτοιου συστήματος. Το είχαμε προβλέψει από την πρώτη στιγμή. Θεωρητικά το 34% των ψήφων θα οδηγούσε στο 100% των εδρών αν εφαρμόζαμε αυτή την κατανομή των ψήφων σε ολόκληρη τη χώρα. Θα υπήρχε αυτή η συνολική στρέβλωση κατανομής των εδρών. Άρα δεν μας εκπλήσει. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε κατά νου γιατί η μουσουλμανική αδελφότητα είχε τόσο υψηλό ποσοστό. Κατά την εποχή του, τη διακυβέρνηση του Μουμπαράκ, η μουσουλμανική αδελφότητα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για να υποστηρίξει τον πληθυσμό ως προς τις κοινωνικές του ανάγκες. Άρα κατά τη στιγμή των εκλογών, κατά τη διενέργεια των εκλογών και με τα μέσα που είχαν, δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το θέμα, με αυτά τα μέσα όμως που διέθηκαν, ανταμείφθηκαν για αυτό που έκαναν κατά τη διακυβέρνηση του Μουμπαράκ, γιατί ήταν η μόνη αντιπολίτευση αν και όχι πολιτικής υφής. Τα είχαν καταφέρει πολύ καλά λοιπόν και είχαν βοηθήσει τον Αιγυπτιακό λαό. Και γι' αυτό και τους επενούμε. Και ανταμείφθηκαν κιόλας. Τώρα πώς διαγράφεται το μέλλον. Καταρχήν συμφωνώ με τον Σάμι όταν μιλά για το ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων, για το ΣΚΑΦ. Ε, δεν είναι πολύ οργανωμένη σκέψη μου όσο μιλώ, θυμάμαι και άλλα. Μην ξεχνάτε τι έγραψε η Λιμπερασιόν ένα χρόνο πριν. Αυτά που θα δούμε στην Αίγυπτο θα είναι ε, μία πλήρης ανατροπή των καταστάσεων. Δηλαδή, ε, θα υπάρχει ε, ψήφος, δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο μία φορά. Αυτό έγραφε η Λιμπεράσιο. Α ελπίσουμε να μην ισχύσει κάτι τέτοιο. Βεβαίως εξαρτάται από τους Αιγύπτιου. Εμείς δεν θέλουμε να δίδουμε μαθήματα σε άλλες χώρες. Κάθε χώρα είναι αυτοκυρίαρχη αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν κάνει ορισμένες υποδείξεις. Έχετε λάβει και στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο μία επιστολή από την Κάθη Άστον και τον Επίτροπο Φίλε για την ε, πολιτική More for More στην, ε, στην πολιτική γειτονίας. Πρόκειται για μία νέα αρχή αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να επιβάλλουμε αρχές στην πολιτική γειτονίας, αλλά θέλουμε να δούμε τις ε, σχέσεις, πώς διαγράφονται και όταν μιλάμε για περισσότερη υποστήριξη σε χώρες, σε γείτονες χώρες, ως προς την ε, υλικοτεχνική αυτή υποστήριξη, ακολουθούμε αυτή την αρχή του more for more. Τώρα ως προς τους ε, δημοσιονομικούς πόρους θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μία προοδευτική ε, υποχώρηση υπάρχει μια παλινοδία ως προς τον τουρισμό. Ξέρουμε ότι οι τουρίστες της ε, Αιγύπτου ανέρχονται στο 30% ε, σε σχέση με πριν από την Επανάσταση. Αυτό είναι λάθος. Δεν θέλω να πω ότι είναι 3%, αλλά δεν καν 30%. Δυστυχώς είναι πολύ χαμηλότερο το ποσοστό του τουρισμού. Έχω έναν φίλο που έχει παντρευτεί μια Πορτογαλίδα και είναι διευθυντή ενός από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του Καΐρου και μου είπε ε, «Μάριο, έχω έξι επισκέπτες στο ε, ξενοδοχείο μου που διαθέτει 700 ε, δωμάτια, δεν θέλω να πω περισσότερα». Δεν θέλω να σας πω, δεν θέλω να φαίνεται ότι δίνω δημοσιότητα και προωθώ ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο παρόλο που είναι πολύ καλό. Μπάς περιπτώσει, ο τουρισμός έχει πέσει δραστικά. 7 με 8 εκατομμύρια Αιγυπτίων που ζουν στο εξωτερικό εμβάζουν χρήματα στην Αίγυπτο. Όμως έχει μειωθεί αυτό το ποσοστό εξαιτίας των γεγονότων της Λιβύης. Αυτή είναι μια πρώτη πραγματικότητα. Και αν λάβετε υπόψη την ανησυχία και την ε, ε, ε, και την αβεβαιότητα που επικρατεί, οι μετανάστες δεν εμβάζουν χρήματα στη χώρα τους. Το ίδιο σημαίνει και στην Πορτογαλία, στην ε, χώρα μου. Αλλά σας παρακαλώ μην το αναφέρετε παράξω. Μία τρίτη, ένα τρίτο θέμα είναι η διόρυγα του Σουέζ, το πέρασμα αυτό, τα, τα δικαιώματα ε, διέλευσης. είναι η μόνη πηγή εσόδων που δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την κατάσταση πριν από την Επανάσταση. Μιλάμε όμως για μια βαθμιαία μείωση εσόδων. Δηλαδή κάθε φορά έχουμε να κάνουμε με λιγότερο από το ημισού του προηγουμένου. Ως προς τις εξαγωγές ε, φυσικού αερίου δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι ο αγωγός που περνάει από την Ιορδανία και το Ισραήλ έχει καταστραφεί. Άρα τα έσοδα από τον αγωγό είναι ανύπαρκτα. Έλεγα στους Αιγύπτους φίλους ότι η Αίγυπτος είναι μία από τις τελευταίες χώρες όπου θα ήθελα να είμαι πολιτικός παρά τα προβλήματά της. Έχει 80 εκατομμύρια ε, πληθυσμό ακολουθεί μία διαδικασία εκδημοκρατισμού. Και επειδή μιλάμε για μία αύξηση, ραγδαία αύξηση και, του, και στον ε, τομέα της, ε, των γεννήσεων, πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε σε ε, σχέδια, προγράμματα υποδομής. επειδή δεν ε, έχετε και ε, μεγάλα έσοδα από το πετρέλαιο, δεν βγαίνουν βαρέλια και βαρέλια κάτω από τη γη. Δεν υπάρχουν ε, έσοδα από την εξόρυξη πετρελαίου. Φοβάμαι λοιπόν ότι στο εγγύς μέλλον οι άνθρωποι θα αρχίσουν να σκέφτονται ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν. Πάλι υπήρχαν επικρίσεις και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη την κατάσταση και οι στρατιωτικές, ε, οι ένοπλες δυνάμεις και οι πολιτικές δυνάμεις, και εδώ αναφέρομαι στη μουσουλμανική αδελφότητα, θα πρέπει να δουν τι κοινωνία θέλουν να χτίσουν μέσω πρόθεσμα τι σύνταγμα θα ε, εκπονήσουν, πώς θα κυρώσουν το σύνταγμα, γιατί θα πρέπει να κυρωθεί το σύνταγμα με δημοψήφισμα, έτσι ώστε ο πληθυσμός να δει σε τι κοινωνία θα ζει. Είμαι πολύ απογοητευμένος αυτή τη στιγμή με την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά τρέφω ελπίδες ότι τα πράγματα θα αλλάξουν ε, κάπως έτσι ώστε να προωθηθεί η ευημερία του Αιγυπτιακού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα που υπογραμμίσατε την πολιτική κατάσταση και τις εξέλιξεις. Θα χρειαστούμε ακόμη 10 λεπτά. Να και ξεκινήσαμε και 15 λεπτά πιο αργά. Τα δικαιούμαστε. Η κυρία Νασίρα Βολό επικεφαλής ε, του Γραφείου Μέση Ανατολής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη δική μας έποψη, θα ήθελα να πω ότι οι αξιολογήσεις και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν στη συζήτηση μας βρίσκουν σύμφωνο. τις συμμεριζόμαστε πολιτική εικόνα ε, θεωρούμε ότι η Αίγυπτος περνάει από μια δύσκολη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης Πολλά ακόμα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως η παραμονή στην ισχύ στην εξουσία των στρατικών, τα στρατιωτικεία που δικάζουν ε, πολίτες ε, και ούτω καθεξής. Ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης είναι η καταστολή βάρος των μη κυβερνητικών οργανώσεων και σε αυτό η ίδια είπατε εκπρόσωπος εξέφρασε τις ανησυχίες της για την κατάσταση αυτή η Υπηρεσία εξωτερική δράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενιαία Η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί πυλώνα της πολιτικής και η κοινωνία των πολιτών είναι, η, είναι ο κινητήρας αυτής της μεταλλαγής. Συντομώ λοιπόν με διάφορους τρόπους, σε διάφορους τόνους από τις αρχές της Αιγύπτου να θέσουν πέρας στο φαινόμενο αυτό, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Επίσης νομοθεσία σχετική με τις ενώσεις προσώπων ε, είναι εν εξελίξη, βρίσκεται σε επεξεργασία και απαιτούμε να προσαρμοστεί στις ε, διεθνείς προδιαγραφές, πράγμα το οποίο θεωρούμε σημασίας. Οι πρεσβείες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κάιρο ενωμένες κινητοποιούνται σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε, μια, ένα ε, μέτωπο ενωμένο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε σχέση με τις ε, Αιγυπτιακές αρχές. Ο Μπερνατρό Λεόν είναι δικός εκπρόσωπος ε, χτες και σήμερα ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά και τα επισήμανα στις Αιγυπτιακές αρχές. Υπάρχουν διάφορες συνεδριάσεις υψηλού επίπεδου με τις ε, αρχές στην Αίγυπτο και πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας σε κάθε επίπεδο. Επίσης, το State Department, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, που επίσης αντιμετωπίζει δυσκολίε ε, και σε σχέση με τις δικές της ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, καταστολή. Ναι, υπάρχουν ευρωπαϊκέ και αμερικανικέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά ταυτόχρονα και τοπικές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις με αποκλειστικά Αιγύπτιους εργαζόμενου που επίση ε, μετώπισαν αυτή την καταστολή, δεν πρέπει να το λησμονούμε. Για τη διαδικασία των ε, εκλογών συμφωνώ ότι εξελίχθηκαν ομαλά, αλλά υπήρξαν κάποια προβλήματα. Δεν μπορούμε βέβαια να αμφισβητήσουμε το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρηση Προετοιμαζόμαστε όμως να αναλάβουμε επαφή με τις αρχές που θα προκύψουν από την διαδικασία αυτή επαφή όπως είπα διότι δεν ήμασταν σε θέση να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία μέσω της ε, αποστολής παρακολούθησης των εκλογών αλλά υποστηρίζουμε τις τοπικές αρχές και έχουμε διπλωματική μονάδα παρατήρηση επιτόπου. Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε εκ του συναγγείς την διαδικασία και το μήνυμα που θέλετε τώρα είναι ότι πρέπει να προχωρήσει προς μια μη στρατιωτική διακυβέρνηση η Αίγυπτος το ταχύτερο δυνατό. Και περιμένουμε τώρα το, το Συμβούλιο των Ενωπών Δυνάμεων να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο θέμα αυτό. για την οικονομία και τελευταία παρατήρηση που ακούστηκε για την επιδείνωση των οικονομικών συνθήκων. Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί τράπεζα επενδύσεων κοιτούν πώς μπορούν να περιορίσουν τις ανάγκες σε χρηματοδότηση. Προσπαθούν οι Αιγυπτιακές Αρχές να διαπραγματευτούν το Εθνικό Ταμείο μια συμφωνία και πάλι εδώ θα πρέπει να ενσωματωθεί και το θέμα της καταστολής εις βάρος μη κυβερνητικών οργανώσεων και γενικότερα το ζήτημα του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και αρχών. Γιατί ναι, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εφαρμόζεται είναι η πολιτική πιο πολλά για πιο πολλά. Αυτή είναι η βασική μας πολιτική. Με τις πολιτικές βέβαια συνέπειες πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη. Ευχαριστώ θερμά, λέει Πρόεδρο. Δύο συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Θέλει κανεί άλλο. Κυρία Μπράντνερ, τη σημειώνω, αλλά πρώτα κυρία Τεκεζέχ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πρώτη παρατήρηση. Θα ήθελα να πω ότι με συγκλονίζουν αυτά που άκουσα για, την, για το Ίδρυμα Denauer και θα ήθελα να προτείνω στους συναδέλφους μια και έχουμε ως κατεπήγον το ανθρωπιστικό ζήτημα στην Αίγυπτο ε, την επόμενη εβδομάδα που πρόκειται να καλύψει τα μάλλον αθλητικού χαρακτήρα αγωνιστικού χαρακτήρα γεγονότα αλλά μια και έχει γίνει δεκτό το ζήτημα αυτό θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε και με μια αναφορά στο Ίδρυμα Denauer. Αυτά. Για δε ε, τα αποτελέσματα είπατε ότι περιμέναμε να επικρατήσουν οι αδελφοί μουσουλμάνοι στο Αλνούρ. Από την... Ε, μάλλον σε σχέση με το Αλνούρ. Αλλά πρέπει να απαντήσω εγώ ότι με μια διαδικασία πολύ δημοκρατική πριν από χρόνια στην Παλαιστίνη και που επικράτησε η Χαμάς ήδη φαινόταν αυτή η τάση που τώρα φαίνεται να γενικεύεται. Και εκεί που πρέπει να πω ότι έχω πραγματικά καταπλαγεί είναι η συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα ποσοστά της Αλνούς. Ε, και θα ήθελα να μου το εξηγήσει γιατί ίσως κάποιος να θυμάται, τον είχαμε πάει στο Σουδάν ε, πέρσι, είχα μείνει στο Βόρειο Σουδάν για αρκετέ εβδομάδες και εκεί γινόταν πολλής λόγος. Φανταζόμουν ότι πρόκειτο για στρατηγική, για ε, πολιτική του Αλβασίρ. Μιλούσαν λοιπόν για ε, μεγάλη άνοδο των σαλαφιστών στο Βόρειο Σουδάν πάντα που έρχονταν με πολύ χρήμα και εξαγόραζαν ψήφους. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν θεωρείτε ότι σε αυτή την σημαντική άνοδο της Αλνούρ στην Αίγυπτο βλέπετε μια αντίστοιχη εξήγηση αντίστοιχο φαινόμενο. Άλλωστε το Σουδάν δεν είναι και πολύ μακριά. Και επίση θα ήθελα να ρωτήσω για να κλείσω εάν έχουμε κάποια ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Καταρχήν βέβαια δεν γνωρίζουμε, αλλά στην ουσία ίσως δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία, αν θέλετε να μου απαντήσετε. Καλώς, ευχαριστώ. Βλέπω κάποιους συναδέλφους που μπαίνουν για την ακρόαση τη σχετική με τη Ρωσία. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά θα αρχίσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Κυρία Ρομέρο Λόπες. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω την ακρόαση αυτή και το ραντεβού μας με το Ίδρυμα Αντενάουερ γιατί όπως είπε και η συνάδελφος ε, Βερονίκ έχουμε να κάνουμε με συμπτώματα μίας γενικότερης κατάστασης δηλαδή μιλάμε για μία ε, κατάσταση συνεχών ε, παλινοδιών. Θα ήθελα να πω προς τον κύριο Σαμί ότι γνωριστήκαμε στη ε, Ρώμη, στην ε, Ένωση, στην Ευρωμεσογειακή Ένωση. Όπως ξέρετε, εγώ προέρχομαι από την Ανδαλουσία και είχα δώσει μεγάλο αγώνα για τις ελευθερίες στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη και αυτό εν μέρη οφείλεται και στο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο ρόλος της μουσουλμανικής αδελφότητας οδηγεί σε αβεβαιότητα, διότι πολλές φορές και σε όλα υπάρχει εποπτεία του στρατού. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μία ε, δημοκρατία αστικού χαρακτήρα όπως θα επιθυμούσαμε. Βλέπουμε ότι παλινοδούμε και οπισθοδρομούμε και αυτό θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος και της ε, μουσουλμανικής αδελφότητας και αυτό αφορά και τα Ισλαμικά κόμματα στη, στο Μαρόκο, στην ε, Τουρκία και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά όλα εξαρτώνται από το πώς θα δράσει η δημοκρατική αντιπολίτευση και πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μία καλώς διαρθρωμένη αντίδραση και αντιπολίτευση έτσι ώστε να αλλάξει το Σύνταγμα πριν από τις προεδρικές, γιατί δεν μπορεί με ένα 70% μουσουλμάνων να ε, ε, οριστεί ένα σύνταγμα το οποίο ανταποκρίνεται στη θέληση του λαού. Θα πρέπει στο μέλλον να αλλάξει. Γι' αυτό η αντιπολίτευση που επιθυμεί δημοκρατία, καθαρή δημοκρατία χωρίς στρατιωτική εποπτεία να ορίσει για, μια, για ένα πραγματικά δημοκρατικό σύνταγμα. Εκεί όπου υπάρχει βία των νέων στην πλατεία Ταχρήρ και αλλού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειρηνικά μέσα να αναγνωριστεί μια πραγματική αντιπολίτευση και ένας εναλλακτικός λόγος σε αυτή τη μουσουλμανική αδελφότητα, χωρίς την εποπτεία του στρατού. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά πρόκειται για μια βραδία διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει καλώς διαρθρωμένη αντιπολίτευση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπράντσινας πολύ σύντομα και θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις και τώρα τον κύριο Γκυρούλη το πολύ σαφή του λόγια. Μια ερώτηση τώρα για τη διαδικασία αυτή της τέξης νέου συντάγματος Φαντάζομαι ότι είτε θα προσδοριστούν κάποιοι βουλευτές που θα συμμετάσχουν στην ε, σύνταξη του νέου κειμένου είτε όχι. Ε, υπάρχει κάποια διαδικασία συγκεκριμένη, σας έχουν ζητήσει βοήθεια, συμβουλές, υποστήριξη, ζητούν προς τα έξω κάποια στήριξη. Η Επιτροπή της Βενετίας ενδεχομένως. και υπάρχει κάποια δυνατότητα, το λέτε κύριε Ντουόρκ, είναι παραδείγμα ότι μπορεί να προχωρήσουν όλα αυτά χωρίς ευρύτερη συμμετοχή. Μπορεί κανείς από εμά να βοηθήσει ώστε να εξελιχθεί η διαδικασία χωρίς να φανεί ότι η συμμετοχή της Δύσης είναι παρέμβαση. Αυτό θα ήθελα, να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο τι συμβαίνει ακριβώς και τι έχει προγραμματιστεί, τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Έχω σοβαρό πρόβλημα χρόνου, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ τον κύριο Σαμί να απαντήσει πολύ σύντομα, τον κύριο Ντουόρκιν επίση πολύ σύντομα. Και γενικά και στην κυρία Μπράντνερ όμως ε, ε, επιμέρους. Κύριε Σάμι, ευχαριστώ. Καταρχάς ε, για τους ε, εργαζομένους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ε, ακτιβιστές καλύτερα, που δεν είναι Αιγύπτιοι, παπιλούνται με πέντε χρόνια φυλακή εάν καταδικαστούν και είναι βέβαιο ότι θα καταδικαστούν σε ένα τουλάχιστον με μέγιστο πέντε χρόνια φυλάξη, εάν, ε, θεωρηθεί ότι έχουν κάνει κάποιες αιτίε δραστηριότητε. Η ΣΚΑΦ τώρα. Η ΣΚΑΦ είναι μια οργάνωση, το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι μια οργάνωση η οποία έχει ζητήσει ε, τη διεθνή συνεργασία σε πρώτη φάση για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία τη καταστολή τη βάρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και ένα από τα πιο σοβαρά, πιο σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει το Κοινοβούλιο σα να επισημάνει στο το Συμβούλιο θα ήταν για την ε, κυρία Μπουνάγκα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πράξει αυτό το Κοινοβούλιο, αλλά όσο ε, ε, ε, ε, εάν υπάρχει δυνατότητα να εγκριθεί αυτή η βίζα της κυρίας Σαμπουνάγκα και των λοιπόν που βρίσκονται στο πλευρό της για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Πρώτη απάντηση. Δεύτερον, για του ελαφιστέ. Ε, πρώτον, το στρατό δεν ψηφίζει, δεν συμμετέχει στι ε, ε, εκλογικέ διαδικασίε. Ξέρω ότι δεν συμβαίνει το ίδιο για το Σουδάν, αλλά στην Αίγυπτο δεν ψηφίζει ο στρατό στι εκλογέ. Πάντω υπάρχει ξεκάθαρα ε, σύνδεσμο μεταξύ σαλαφιστών, μουσουλμάνων αδελφών και αδελφών μουσουλμάνων και στρατού. Στην Αίγυπτο είναι ξεκάθαρο. Επίσης, ακούστηκε νωρίτερα ότι η Αίγυπτος έχει ορμή, έχει όθηση. Ναι, αλλά και ο λαός έχει πολύ φυσικό αέριο. Ωστόσο, ο λαό έχει πρόβλημα, πρόβλημα ω προ την προμήθεια σε φυσικό αέριο. Δηλαδή, φτάνει το φυσικό αέριο τελικά στα σπίτια του κόσμου. Έτσι λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι σαλαφιστέ έχουν τη δυνατότητα τη άμεση πρόσβαση στι πηγέ του φυσικού αερίου και το φέρνουν οι ίδιοι στα σπίτια του, των πολιτών και τα προσφέρουν, προσφέρουν τις μπουκάλες του αερίου με πολύ χαμηλές τιμές εξασφαλίζοντας έτσι και την ψήφο του κόσμου. Έχουμε βέβαια μια διαδικασία συνταγματική. Ε, υπάρχει περίπτωση, όπω είπατε, να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σα λέω δεν πρόκειται να βοηθήσει παρά μόνο του Ισλαμιστέ κανέναν άλλον. Ε. Και το μόνο που μπορώ να συστήνω είναι όταν κοιτάτε, όταν μελετάτε την Αίγυπτο, δείτε την σαν μια Αλγερία του 90, αλλά και σαν μια, Τουρκία του 80, τη του 80. Είναι ένα μείγμα των δύο αυτών κρατών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ τους πάντες ε, θερμά για την παρουσία τους και τις παρουσίες τους. Θα συνεχίσουμε και με, τα, και με το κατεπήγον που έχουμε την επόμενη εβδομάδα, αλλά και με την παρακολούθηση της κατάστασης. Το επόμενο θέμα είναι και κλεισμένο των θυρών. Και παρακαλώ όποιος είναι να έρθει να συζητήσουμε για το θέμα της, της Ρωσίας όποιος δεν δικαιούται να αποχωρήσει.